Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Άρχεται η συνεδρίαση τη Επιτροπή μας. Βλέπετε εδώ νέα πρόσωπα. Και αυτό γιατί βεβαίω δεν υπήρχε κανείς άλλος από το Προεδρείο, οπότε ζήτησαν από εμένα να προεδρεύσω μια που είμαι ο πρεσβύτερος. Οπότε έτσι και έγινε. Έχετε όλη την ημερήσια διάταξη. Έχετε σχόλια. Αν όχι εγκρίνεται, περνάμε στο δεύτερο σημείο ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Πρέπει να σας πω πως έχουμε τον κύριο Σβέτιτς, ένα νέο υπάλληλο στην γραμματεία, τον οποίο καλωσορίζω στην Επιτροπή μας. Ναι, ναι, είναι από την Κροατία επίσης να σας πω. Οπότε έχει και κάποια, κάποιο όνομα να διατηρήσει. Έχουμε λοιπόν βουλγαρικά, ελληνικά μεταξύ πολλών άλλων. Υπάρχει κάποιος παραπονεμένος που θεωρεί πως δεν υπάρχει γλώσσα του. Όχι, ούτε αυτό. Οπότε Πρέπει επίσης να σας προειδοποιήσω πως ό,τι πείτε θα το παρακολουθήσει όλος ο πλανήτης γιατί μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Σημείο 3. Της ημερήσιας διάταξης. Πρέπει να εγκρίνετε τα πρακτικά των συνεδριάσεων 4 και 5 Νοεμβρίου, 7 Νοεμβρίου, 14 Νοεμβρίου και 25 και 26 Νοεμβρίου. Σχόλια για τα πρακτικά. Όχι. Οπότε εγκρίνονται. Περνάμε στο σημείο 4. Απαλλαγή 2012. Έχουμε εδώ πέρα τον Επίτροπο Χάν, τον αρμόδιο για την περιφερειακή ανάπτυξη και το αρμόδιο μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου, τον κύριο Γκέτεν. Καλωσορίζω και τους δύο λοιπόν και θα δώσω λόγο στον κύριο Πίπερ τον εισηγητή μας. Ναι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητό μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είναι νομίζω μια αποφασιστική, σημαντική συνεδρίαση στο πλαίσιο της απαλλαγής και η ανακοίνωση την οποία ε, είχα βγάλει εγώ μαζί με τους άλλους και οδησυγητές και απευθυνόταν προς τον κύριο Μπαρόζο. Ε, ελπίζαμε πως θα έχει απαντηθεί, πως θα έχει υπάρξει κάποια αντίδραση από πλευράς Κομισιόν. Οπότε τουλάχιστον έχουμε κάτι και γι' αυτό σας ευχαριστώ τώρα. Να αναφερθώ στα ερωτήματα τα οποία απαντήθηκαν γέρος. Θεωρώ πως ε, τα περισσότερα απαντήθηκαν ικανοποιητικά. Κάποια πράγματα βεβαίως ήταν στα ελληνικά, ε, με τα οποία ακόμη παλεύουμε, αλλά αναμένουμε κάποιες απαντήσεις. Θα τα δουν αυτά βεβαίως για τις λεπτομέρειες οι συντονιστές μας. δεν ξέρω αν το ελεγκτικό συνέδριο είναι σε θέση να κάνει κάποια δήλωση, κύριε Ρέτεν, για την ανακοίνωση αυτή. Ωραία, ωραία. Αλλά θα ήθελα πρώτα να αναφερθώ στο βασικό θέμα που μας απασχολεί, τι γίνεται δηλαδή με τα διαρθρωτικά ταμεία. Όλοι ξέρουμε πως τα λάθη είναι ανθρώπινα. Αλλά όταν γίνονται συνεχώς τα ίδια λάθη, τότε νομίζω κάποια στιγμή πρέπει να βρούμε και τον φταίχτη, να τον κατονομάσουμε. Δηλαδή θα κάνω μια παρομοίωση με τον κοκ. Άμα συνεχώς παραβιάζω τον κόκ, κάποια στιγμή χάνω το δίπλωμά μου. Και πάντα τα ε, ίδιες πηγές είναι ε, των σφαλμάτων, δηλαδή οι δημόσιες προμήθειες και οι μη επιλέξιμες δαπάνες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτές. Και πάντα τα ιδια κρατη καράτη-μέλη, τα οποία κάνουν κατά κύριο λόγο τα σφάλματα. Είναι λοιπόν μη ικανοποιητική κατάσταση να απαντάμε και να λένε, να μας απαντάνε και να λένε του χρόνου καλύτερα ή στην επόμενη προγραμματική περίοδο καλύτερα. Ε, τα ίδια γίνονται τα τελευταία 15-17 χρόνια. Αλλά θέλουμε κάποια στιγμή να γίνει κάποια ουσιαστική πρόοδος εδώ πέρα. που έρχονται και ευρωεκλογέ και ως κοινοβούλιο αναμένουμε και βεβαίως αναμένουν και από εμάς να δούμε το θέμα με κριτική διάθεση, να μην προστατεύουμε κανέναν, να εκπληρώσουμε την εντολή μας για διαφάνεια βεβαίως παρακολουθούμε τη διαδικασία και έχουμε ακόμα κάποιες ερωτήσεις τώρα. Να έρθω. Λίγο πιο πολύ στην ουσία. Ένα θέμα είναι η γεωργική ανάπτυξη. Δεν είναι το σημερινό θέμα, αλλά βεβαίως εκεί πέρα έχουν μείνει πιο πολλά ανοιχτά ερωτήματα από αυτά τα οποία απαντήθηκαν. Μετά, διαρθώτικα ταμεία. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα ποια είναι αυτή η προσέγγιση με βάση την ανάλυση κινδύνου. Από πότε, δηλαδή από ποιο σημείο θα αρχίσει να παρεμβαίνει η Κομισιόν. Έχουν εντύπωση πως εδώ υπάρχει κάποια διακριτική ευχέρεια την οποία δεν μπορεί να παρακολουθήσει κάποιος που είναι απ' έξω. Δηλαδή, σε ποιες χώρες, με, ποια, με ποιους δειγματολογικούς ελέγχους και με ποιο όριο αποφασίζετε να παρέμβετε. Κύριε Επίτροπε, αυτό ήταν το βασικό αντικείμενο της επιστολής μας προς τον κύριο Μπαρόζο. Θέλουμε έναν αυτοματισμό, τον οποίο να μπορούμε να παρακολουθήσουμε και εμείς ως κοινοβούλιο. Και να μην αφήνουμε περιθώρια, όπως είπα, διακριτικής ευκαιρία στην Κομισιόν. Ποια είναι τα όρια και πώς μπορούμε εμείς να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία. Και το άλλο το οποίο οπωσδήποτε πρέπει να γίνει και μας είπατε ότι θα γίνει, τι κάνουμε με τους υπότροπους. Είπατε πως θα υπάρξει κάποια πράξη κατεξιοδότηση κάποιο, κάποια σχετική πρόβλεψη. Μας είπατε πως το Φεβρουάριο θα έχουμε κάτι σχετικό, το οποίο αναμένουμε. Θα πάει το σχέδιο της έκθεσής μου τότε για μετάφραση, οπότε υπάρχει ακόμα χρόνος ε, να το δούμε, αλλά πραγματικά πρέπει αυτό να είναι το επόμενο βήμα. Αυτό αναμένουμε από τον Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την ομάδα του. Αυτά τα υπόλοιπα θα τα αφήσω, θα τα πούν και οι συνάδελφοι. Νομίζω αρκεί μια δική μου δήλωση επί της αρχής και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πάρα πολύ την βάση που είχαμε για να αποστείλουμε απευθείας μία επιστολή στον πρόεδρο της Κομισιόν. Μπορεί σε κάποια σημεία να μην συμφωνούμε απολύτως με το ελεγκτικό συνέδριο, αλλά αυτά τα οποία νομίζω μας έδωσε ως στοιχεία είναι πάρα πολύ πολύτιμα. Δεν θα χαλαρώσουμε, θα παραμένουμε αυτά τα οποία μας υποσχεθήκατε και όσον αφορά τις εκθέσεις αναχώρα για τα διαρθρωτικά ταμεία, για τη γεωργία. Αλλιώς ε, αυτά τα οποία μας έδωσε το ελεγκτικό συνέδριο στην άλυση του είναι πάρα πολύ ικανοποιητικά. Αυτά λοιπόν ως δικές μας εισαγωγικές ε, παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο τώρα έχει ο κύριος Γκρέτε με το ελεγκτικό συνέδριο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής ε, και το Κοινοβούλιο για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν την προηγούμενη εβδομάδα για την ανανέωση της εντολής μου. Μπορώ να σας υποσχεθώ πώς θα συνεργαστώ με το Κοινοβούλιο, πώς γνωρίζω πως το Κοινοβούλιο είναι ο εντολέας μας και εργαζόμαστε για τον Ευρωπαίο πολίτη, οπότε σας ευχαριστώ ακόμη μια φορά για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε. Δεύτερον, να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Πίπερ. Ε, βιάστηκα και είπα πως το ελεγκτικό συνέδριο θα μπορούσε ήδη σήμερα να τοποθετηθεί επί της έκθεσης της Κομισιόν. Σήμερα την λάβαμε, επισήμως δεν την έχουμε λάβει, δυστυχώς λοιπόν θα πρέπει να επιδείξετε κάποια υπομονή πριν τοποθετηθούμε συλλογικά. Ναι, ναι, βεβαίως, αλλά πρέπει να ρωτήσω για του υπόλοιπου 27 συναδέλφου. Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι σήμερα που μπορώ να σας αναφέρω τα αποτελέσματα του κεφαλαίου 5 τη ετήσια έκθεση Συνεδρίου για το 2012. Εκεί πέρα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για την περιφερειακή πολιτική ενέργεια μεταφορά και προπολογισμό. Το κεφάλαιο 5 καλύπτει συνολικά πληρωμές γύρω στα 41 δισεκατομμύρια ευρώ και η περιφερειακή πολιτική είναι 96% αυτής της, ε, αυτών των ποσών. Μιλάμε για πάνω από 180 πληρωμές ε, και καταλήξαμε πως το ποσοστό σφάλματος ε, για ε, περιφερειακή πολιτική ενέργεια και μεταφορές βρίσκεται μεταξύ 3,7 και 9,9%. 6,8% είναι το πιο μεγάλο πιθανό ποσοστό σφάλματος. Είμαστε δηλαδή πάνω από το ποσοστό σημαντικότητας του 2% όμως είναι σημαντικά χαμηλότερο από το ποσοστά σφάλματος που είχαμε για την περίοδο 2000-2006. Πέρα από το εκτιμόμενο ποσοστό σφάλματος υπολογίσαμε έναν άλλο σημαντικό δείκτη που αφορά την εφαρμογή του προϋπολογισμού. Πρόκειται για την συχνότητα σφαλμάτων. Ο δείκτης αυτός μας δείχνει ποιο ποσοστό των συναλλαγών που εξετάσαμε επηρεάστηκε από οποιοδήποτε είδος σφάλματος σημαντικού ή λιγότερο σημαντικού. Στον τομέα αυτών λοιπόν 88 από 180 συναλλαγές που ελέγξαμε είχαν σφάλματα. Δηλαδή έχουμε ένα 49% των συναλλαγών που ελέγξαμε το 2012. Λίγο παραπάνω από τις μισές ε, συναλλαγές που είχαν σφάλματα είχαμε επαρκείς πληροφορίες ε, και θα έπρεπε να τα ε, έχουν ανοιχνεύσει οι αρχές των κρατών μελών πριν βεβαιώσουν τις δαπάνες προς την Κομισιόν. Τα περισσότερα σφάλματα που βρήκαμε οφείλονται σε μη συμμόρφωση με του κανόνες για τι δημόσιε προμήθειε. Τα λοιπά αφορούν προβλήματα επιλεξιμότητας και το μη σεβασμό των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. Πριν συνεχίσω, θα ήθελα να τονίσω πως σφάλμα δεν σημαίνει οπωσδήποτε σπατάλη ή απάτη να αναφερθώ πρώτα απ' όλα στα σφάλματα που αφορούν τις δημόσιες προμήθειες. Όπως και σε προηγούμενα χρόνια, το ελεγκτικό συνέδριο βρήκε πως ο μη σεβασμός των κανόνων ήταν η μεγαλύτερη πηγή παρατυπιών. Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως σφάλμα δεν σημαίνει οπωσδήποτε πως το ίδιο το έργο δεν παραδόθηκε ως όφιλε. Επίσης θα ήθελα να επισημάνω πως Λόγω της σημασίας των δημοσίων προμηθειών, το ελεγκτικό συνέδριο σκοπεύει να αναλάβει έναν έλεγχο του θέματος. Δεύτερον, λίγα λόγια για τα λάθη επιλεξιμότητας, όπου θεωρούμε πως οι κανόνες επιλεξιμότητας δεν έγιναν πλήρως σεβαστοί. Τα ίδια τα κράτη-μέλη όρισαν αυτούς τους κανόνες, όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών δηλαδή. Τρίτον, τα σφάλματα που αφορούν τη μη συμμόρφωση με κανόνες ε, για τις κρατικές ενισχύσεις. Εκεί πέρα διασφαλίζεται πως οι παρεμβάσεις των κρατών μελών δεν διαστευλώνουν τον ανταγωνισμό. Ως βασικός κανόνας που προκύπτει από την ε, συνθήκη, οι κρατικές ενισχύσεις δεν είναι νόμες εκτός εάν επιτρέπονται ρητός. Αυτό μπορεί να προκύπτει είτε από την ίδια τη συνθήκη, από κανονισμό ε, όταν μιλάμε για μικρά ποσά ή από συγκεκριμένες αποφάσεις της Κομισιόν μετά από την εξέταση της συμβατότητας της συγκεκριμένης ενίσχυσης με την εσωτερική αγορά. Το κεφάλαιο 5 ε, δίνει ένα παράδειγμα. Στην περίπτωση ενός έργου που αφορούσε λιμενικές εγκαταστάσεις, η ενίσχυση ήταν κρατική ενίσχυση, αλλά δεν ειδοποιήθηκε η Κομισιόν και άρα δεν είχε ε, αξιολογηθεί η συμβατότητα με την εσωτερική αγορά. Επιπλέον θα ήθελα να αναφερθώ στο πώς το ελεγκτικό συνέδριο έλαβε υπόψη τις δημοσιονομικές διορθώσεις το 2012. Πριν συνεχίσω να τονίσω πως το συνέδριο είναι υποχρεωμένο στην ετήσια έκθεση να αναφέρει το εάν είναι νόμιμες και κανονικές οι δαπάνες και οι Κομισιόν είναι υποχρεωμένο να προστατεύσει τα οικονομικά συμφέροντα της κοινότητας. Η προσέγγιση του συνεδρίου και της ε, Κομισιόν είναι διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές. Οι δημοσιονομικές διορθώσεις που επιβάλλει είτε η Κομισιόν είτε οι αρχές των κρατών μελών και που έχουν οδηγήσει σε συγκεκριμένες διορθώσεις δαπανών ή επιστροφή ποσών μείωσαν το ποσοστό σφάλματος αφενός για το 2012 αφετέρου οι καταποκοπήν διορθώσεις που δεν αφαιρούν τις μη κανονικές δαπάνες από την δήλωση στο επίπεδο του έργου δεν επηρεάζουν το ποσοστό σφάλματος που υπολογίζει το συνέδριο. Δηλαδή σε άλλες περιπτώσεις. Σε περιπτώσεις όπου ε, το δικαστήριο, το ελεγκτικό συνέδριο θεωρεί ότι υπάρχει σφάλμα, αλλά δημοσιονομική διόρθωση έχει ήδη επιβληθεί σε επίπεδο έργου, τότε το σφάλμα δεν ε, συνυπολογίζεται στο ποσοστό σφάλματος. Αυτό συνέβη για πολλές συναλλαγές που ελέγχθηκαν το 2012 όπως περιγράφονται στο 1.3 και στην παράγραφο 1.33 του κεφαλαίου 1 της ετήσιας έκθεσης. Τέλος, σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα των συστημάτων, ε, εστιάζουν όπως και σε προηγούμενα έργα στο ρόλο που παίζουν οι ελεγκτικές αρχές των κρατών μελών και στη δουλειά που κάνει η Κομισιόν για να υποπτεύσει αυτό το έργο. Η ευθύνη για τον έλεγχο των περιφερειακών δαπανών ε, την επιμερίζονται τα κράτη-μέλη μας με την Κομισιόν. Σε ό,τι αφορά τις ελεκτικές αρχές το 2012, το συνέδριο αξιολόγησε 4 από 112 τέσσερις αρχές που έχουν τα κράτη-μέλη συνολικά. Και καταλήξαμε ότι μία από τις τέσσερις ήταν αποτελεσματική και οι υπόλοιπες τρει ήταν μερικώς αποτελεσματικός. Το συνέδριο βρήκε αδυναμίες στον τρόπο που οι ελεγκτικές αρχές διενεργούν τους ελέγχου και αναφέρουν τα αποτελέσματα. Δεύτερον, το συνέδριο βρήκε αδυναμίε στη δουλειά που, κάνουν, που έκανε η Κομισιόν σε ό,τι αφορά την, ε, τον εποπτικό τη ρόλο στις ε, ελεγκτικές αρχέ λόγω τη ανεπαρκού πληροφορία που δίδεται προς την Κομισιόν όταν ε, κάνει τη δουλειά της. Περισσότερες πληροφορίες ε, για αυτό το θέμα μπορούν να βρεθούν στην ειδική έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Καταγράφοντας τους ελέγχους και τη δουλειά που κάνει η Κομισιόν εποπτεύοντας τις εθνικές Ελεκτικές αρχές» ε, που θα δημοσιευθεί ως ο Νούμπο. Κύριε Σιγητά, αγαπητοί βουλευτές, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Ε, υπάρχει και ένα άλλο μέλος του ελεκτικού συναδρίου ε, παρόν. Εσείς είσαστε ειδικό για τις δημόσιες προμήθειες. Κύριε Λαζάρο, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι υπεύθυνο για το κεφάλαιο 5 από το 2013 και μετά όμως. Δεν έχω να προσθέσω λοιπόν τίποτα για το θέμα αυτό. Μια και ο συνάδελφος όμως ανέφερε κάποια πράγματα, θα ελέγξω τις δημόσιες προμήθειες, έχω αυτό το, αυτή την πρόθεση, όπως είπα στις 5 Νοεμβρίου στην ε, Οικονομική Επιτροπή του Κοινοβουλίου. Θα ξεκινήσουμε έναν έλεγχο επιδόσεων για τις δημόσιες προμήθειες κάποια στιγμή το Μάρτιο ή Απρίλιο του 2014. Ήταν πολύ χρήσιμο που ανταλλάξαμε απόψεις με τα μέλη της ε, Οικονομικής Επιτροπής του Κοινοβουλίου για να δω ποιες είναι οι συγκεκριμένες ανησυχίες τους. Ανταλλάξαμε απόψεις φυσικά και με την Κομισιόν και θα ξεκινήσουμε τις, ε, τους ελέγχους επιδόσεων με ένα σεμινάριο brainstorming στις 29 Ιανουαρίου που θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου, στα γραφεία του Ελεκτικού Συνεδρίου, με ομιλητές από την Κομισιόν, και εμπειρογνώμονες για τα θέματα δημοσίων προμηθειών και ελπίζουμε η ανταλλαγή απόψεων αυτή στο σεμινάριο να μας βοηθήσει περισσότερο, ούτω ώστε να είμαστε πιο εστιασμένοι στις, στους ελέγχους που θα διενεργήσουμε για τις επιδόσεις ε, στις δημόσιες προμήθειες. Ο Επίτροπος έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Γκρέιτεν για την πολύ ισορροπημένη απεικόνηση της περιφερειακής πολιτικής στην ετήσια έκθεση. Για τέταρτη φορά έχουμε μικρότερο ποσοστό σφάλματος από την περίοδο 2006-2008. Ε, αναφερθήκατε στο ότι δεν υπήρξε εδώ πέρα κάποια συνέχεια. Θέλω λοιπόν να σας πω πως βλέπουμε σαφώς την διαφορά μεταξύ των ε, διαφορετικών περιόδων και αυτό το λέω γιατί το ελεγκτικό συνέδριο το 2012 διαπίστωσε μία μικρή αύξηση του ποσοστού σφάλματος. Νομίζω πως ε, στην εφαρμογή των ε, προγραμμάτων μας ε, θα παραμείνει κάπου ένα ποσοστό σφάλματος και αυτό οφείλεται βεβαίως και στην λογική πολυετών προγραμμάτων και στην πολυπλοκότητά τους και τελικά σχετίζεται και με τον ε, κανονισμό. Δεν μπορούμε να, να αγνοήσουμε τελείως τους κανονισμούς μας μαθαίνουμε το μάθημά μας, αντλούμε τα διδάγματα που πρέπει και οπωσδήποτε οι συστάσεις σας εφαρμόζονται στην επόμενη περίοδο. Θα δείτε πως πάρα πολλές έχουν εφαρμοστεί και βεβαίως ε, χρειάζεται και χρόνος για να φανούν τα αποτελέσματα. Συνολικά, αν δούμε τα νούμερα, βλέπουμε μία βεβαίωση μιας ε, θετικής ε, τάσης ο πρόεδρος, ο κύριος ε, Καλντέρα, νομίζω το επιβεβαίωσε εδώ πέρα στην Επιτροπή και νομίζω αυτό οφείλεται και στη βελτίωση του νομικού πλαισίου. Και πέρα από το νομικό πλαίσιο, εξίσου σημαντικό είναι και η συνεπής ε, χρήση και εφαρμογή του. Η Κομισιόν σήμερα ελέγχει ένεργα τα συστήματα διοίκησης και ελέγχου των ε, κρατών μελών και θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε κάποια παραδείγματα. Πρώτον, ε, χρησιμοποιούμε συστηματικά διασταυρώσεις ε, αριθμών και αναλύσεις στοιχείων και εκεί πέρα προκύπτουν κάποια προβλήματα. Το 2012 είχαμε πληρωμές 184 εκατομμυρίων ε, τα οποία ε, αναλύθηκαν 175, σε 175 θα ξεκίνησε μια διαδικασία επιστολής και 13 προγράμματα σε Ισπανία, Ιταλία και Εστονία ξεκινήσαμε αναστολές ε, πληρωμών. Είχαμε επίσης σε 24 από αυτά την διακοπή των πληρωμών και άρα το 2012 μπορούσαμε να επαναλάβουμε τις πληρωμές περισσότερα από τα μισά από αυτά τα προγράμματα. Βλέπουμε λοιπόν πως οι διαχειριστικές αρχές εφάρμοσαν τα μέτρα τα οποία συστήσαμε και άρα η αναστολή των πληρωμών είναι πάρα πολύ σημαντικό μέτρο στην τρέχουσα περίοδο. το 2014 πάμε ένα βήμα παραπάνω. Έχουμε καθαρές δημοσιονομικές διορθώσεις, οι οποίες όμως θα γίνονται κάπως αργότερα. Δεύτερον, δεν διασφαλίζουμε μόνο πως θα εκλείψουν οι συγκεκριμένες πηγές φαλμάτων, αλλά πηγαίνουμε και στο παρελθόν και ε, επιβάλλουμε διορθώσεις. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2013 μόνο με βάση τους ελέγχους της Κομισιόν είχαμε διορθώσεις ύψους σχεδόν ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Τα κράτη-μέλη τα ίδια μας επεσήμαναν ε, διορθώσεις 1,3 ε, δισεκατομμυρίων ευρώ και οι οποίες έγιναν και κατά αποκοπήν και νομίζω πως έτσι διασφαλίζουμε τα οικονομικά συμφέροντα της ε, κοινότητας χωρίς να χρειάζεται να γίνουν ε, διαφορετική έλεγχοι σε χιλιάδες μεμονωμένα έργα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να φροντίζουμε για την ομαλή λειτουργία του συστήματος. Ε, οι καταποκοπήν διορθώσεις παραμένουν ένα σημαντικό μέσο και βεβαίως έχουν και έναν αποτρεπτικό χαρακτήρα. Εδώ πέρα θα ήθελα να αναφέρω και ο συνάδελφός μου ο κύριος Σέμετα το έχει ήδη πει πως το συνέδριο δεν έλαβε υπόψη τις καταποκοπήν αυτές διορθώσεις όσον αφορά το ποσοστό των σφαλμάτων. Όλα αυτά βασίζονται στους κανονισμούς μας. Ο Γενικός Κανονισμός το άρθρο 99 παράγραφος 2 αναφέρει ξεκάθαρα πως υπάρχει δυνατότητα επιβολής τέτοιων ε, κατά αποκοπήν ε, διορθώσεων και επίσης το άρθρο 145 παραγραφός 1. Εκεί πέρα καλύπτεται ο οικονομικός κίνδυνος σφαλμάτων έπαρκος, προστατεύεται ο κοινοτικός προϋπολογισμός και ο Ευρωπαίος φορολογούμενος και επίσης δίνει την δυνατότητα συγκεκριμένης εφαρμογής ε, στα προγράμματα. Είμαι λοιπόν Πεπισμένο πως το ελεγκτικό συνέδριο έπρεπε να έχει λάβει υπόψη και αυτόν τον μηχανισμό και άρα ο υπολογισμός του σφάλματος θα ήταν 0,8% ε, χαμηλότερος. Θα ήταν δηλαδή ακριβώς στο 6% και άρα στο ίδιο επίπεδο με το 2012. Άρα, εδώ πέρα θεωρώ πως ε, συμφωνούμε με τους εκπροσώπους ε, του ελεγκτικού συνεδρίου. Αναφέρθηκε στην παρουσίαση της έκθεσης πως οι προσπάθειες της Κομισιόν για να προστατεύσει τον ε, κοινοτικό προπολογισμό αξιολογούνται θετικά και μέσω των καταποκοπήν διορθώσεων και θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η πορεία. Κάτι το οποίο βεβαίως ε, ήδη αποφασίσατε και εσείς ε, κυρίες και κύριοι βουλευτές ε, στους νέους κανονισμούς για την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο. Θα ήθελα στο πλαίσιο αυτό να αφερθώ στις εθνικές και περιφερειακές ελεγκτικές αρχές. Είναι σημαντική εταίρη και βασικό κομμάτι του μηχανισμού ελέγχου. Πρέπει να λειτουργούν αξιόπιστα. Εμείς ε, στην εποπτική μας λειτουργία επικεντρωνόμαστε κυρίως στη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας τους. Από το 2009 το κάνουμε αυτό συστηματικά, ελέγχουμε ποια είναι τα αποτελέσματά τους, ποιος είναι ο τρόπος λειτουργίας, ποια είναι η μεθοδός τους. Ε, έχουμε κάνει γύρω στους 200 επιτόπιους ελέγχους ε, και έχουμε ελέγξει γύρω στις 147 τέτοιες αρχές δηλαδή σχεδόν το σύνολό τους και τα αποτελέσματα δείχνουν πως μπορούμε να βασιστούμε επάνω τους. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων βεβαίως μπορούν να βελτιώσουν τη λειτουργία τους. Κατά την άποψη την δική μου και των υπηρεσιών μου, δύο πράγματα έχουν μεγάλη σημασία. Επάρκεια του προσωπικού και λειτουργική ανεξαρτησία. Η ετήσια έκθεση των ελεγκτικών αρχών είναι σημαντικό κομμάτι της ε, αξιόπιστης λειτουργίας. Το 2012 ε, μπορούσαμε να βασιστούμε σε ένα 89% των αναφορών που μας έγιναν. Δύο τρίτα δε των ε, σφαλμάτων που εντοπίστηκαν οφείλονται ακριβώς στις εθνικές ελεγκτικές αρχές. Άρα θα έλεγα πως το σύστημα λειτουργεί. Και καταλήγουν και αυτές ε, σε παρόμοια συμπεράσματα σε, ε, με εμάς. αλλά ανησυχώ για το ότι πάνω από το μισό των σφαλμάτων που εντόπισε το ελεγκτικό συνέδριο θα έπρεπε να έχουν ανακαλυφθεί από τις Εθνικές Ελεγκτικές Αρχές πριν μάλιστα αποσταλούν τα στοιχεία στην Κομισιόν. Οι αριθμοί δείχνουν πως ε, δεν λειτουργούν παντού αξιόπιστα τα συστήματα ελέγχου. Τα συστήματα ελέγχου μπορούν να λειτουργήσουν μόνο εάν λειτουργούν σωστά στα κράτη-μέλη και ακριβώς αυτό το πρώτο επίπεδο ελέγχου είναι το σημαντικό που πρέπει να βελτιωθεί. Ήδη από την συζήτηση για την απαλλαγή του 2011 έλαβα το μήνυμα πως θέλετε έναν μηχανισμό με ισχυρότερες κυρώσεις, με πιο αποτρεπτικό χαρακτήρα και με διορθώσεις οι οποίες θα οδηγούν πραγματικά σε ε, μείωση των διαθέσιμων ποσών. Πραγματικά θα το έχουμε αυτό, θα οδηγηθούμε στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο σε πραγματικές ε, ουσιαστικές δημοσιονομικές διορθώσεις. Έχουμε ενισχύσει επίσης την διαδικασία στο πλαίσιο του ελεγκτικού συνεδρίου και θα μπορέσουμε να ανοιχνεύουμε και να διορθώνουμε λάδι πριν οδηγηθούν σε αιτήσει πληρωμής από την Κομισιόν. Και στην περίπτωση στην οποία έχουν αποσταλεί ε, αιτήσει πληρωμής στην Κομισιόν χωρίς να έχουν ε, γίνει αντιληπτά λάθη θα επιβληθούν καθαρές διορθώσεις. Εδώ λοιπόν η Κομισιόν δεν θα έχει κανένα περιθώριο ελεγμών, καμία διακριτική ευχέρεια. Θα ήθελα επίσης ε, να ευχαριστήσω και τους και οδησηγητές για την θετική τους ε, αντίδραση. Ήδη την προηγούμενη Παρασκευή εξέδωσε Κομισιόν μια ανακοίνωση και περιέχεται εκεί πέρα μία σύνοψη του μηχανισμού των καθαρών διορθώσεων από το 2014 και είμαι σίγουρος πως ε, η ανακοίνωση αυτή απαντάει σε πολλές από τις ερωτήσεις σας. Η πολιτική περιφερειακή είναι μια πολιτική κλειδί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχει πόρους για επενδύσεις ε, οι οποίες οδηγούν σε ανάπτυξη και δουλειές, ενισχύει την περιφερειακή συνοχή και ειδικά σε καιρούς κρίσης ακριβώς αυτές οι επενδύσεις στην πραγματική οικονομία έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Το νομικό πλαίσιο για την επόμενη προγραμματική περίοδο έχει στόχο να διαμορφώσει την πολιτική μας πιο απλή, πιο αποτελεσματική και πιο εστιασμένη, αλλά και πιο συνεπή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Θα ε, φροντίσουμε επίσης να έχουμε σαφείς μετρήσιμους στόχους και θα ενισχύσουμε βεβαίως ε, την χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θα ενισχυθεί και η λογοθεσία των κρατών μελών. Κύριε και κύριοι, για να έχουμε βελτιώσεις στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής απαιτείται στενή συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων εθνικών, περιφερειακών και ευρωπαϊκών αρχών τα κράτη-μέλη προσεχώς θα δίνουν περισσότερο λόγο για το πώς διαχειρίζονται τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Η στήριξη της Επιτροπής σας και η δουλειά του ελεγκτικού συνεδρίου νομίζω είναι πολύτιμες και θα είναι και αποφασιστικές στην συνέχεια. Η Κομισιόν θα συνεχίσει να εποπτεύει την κατάσταση στα κρατη για να ε, βοηθήσει και τους πολίτες της περιφέρειας οι οποίοι ταυτόχρονα είναι και φορολογούμενοι Ευρωπαίοι. Σας ευχαριστώ κύριε Επιτροπέ. Ξεκινάει τώρα η συζήτηση. Τρεις ευρωβουλευτές θέλουν να μιλήσουν. Ο κύριος Ρούμπικ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη. Από την πρώτη παρέμβαση του εισηγητή κατάλαβα ότι ήθελε να κάνει κάποιες, κάποια σχόλια μετά την παρέμβαση του Επιτρόπου. Μετά εσείς λοιπόν. Ε, εντάξει κύριε Πρόεδρε. Τρεις ερωτήσεις έχω. Πρώτον, θεωρώ πως η πρόγνωση ε, για το τι θα γίνει από εδώ και μπρος είναι ακούγεται πιστική αλλά το ερώτημα το οποίο έθεσα στην αρχή για τα κριτήρια της ε, αξιολόγησης κινδύνου και της εντονότερης ε, αξιολόγησης υπάρχει κάποιος αυτοματισμός μπορούμε να τον παρακολουθήσουμε και εμείς ως εξωτερικοί δεν το απαντήσατε και Για τον Φεβρουάριο μας έχετε υποσχεθεί ένα νομοθετικό πακέτο. Εκεί πέρα τι έμφαση θα δώσετε στους υπότροπους, όπως είπα. Να μπορείτε να μου πείτε τι προθέσεις έχει η Κομισιόν. Μετά, ένα άλλο ερώτημα για τις δημόσιες προμήθειες. Και εδώ πέρα, εδώ και πολλά χρόνια, έχουμε κάποια προβλήματα, συνεχώς τα ίδια. Υπάρχει μια ετήσια έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς για τις ε, δημόσιες προμήθειες και νομίζω το είδε και η Γενική Διεύθυνση Ρέγγιο. Υπάρχει ένα σχέδιο δράσης πολλών γενικών διευθύνσεων για τις δημόσιες προμήθειες. Συγκεκριμένα, ποιε θα είναι οι βελτιώσεις στον τομέα των δημοσίων προμηθειών στο μέλλον και τι κάνετε συγκεκριμένα στις χώρες που έχουν αυτή την ενδιάμεση διοίκηση όπως η Γερμανία. Δηλαδή, πέραν από την Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία, σε ομοσπονδιακές χώρες, όπως και η Ισπανία. Τι θα αλλάξει συγκεκριμένα. Και κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ επίκαιρο τώρα, θα κάνετε αυτές τις συμφωνίες ε, εταιρική σχέση και θα ελέγξετε τα επιχειρησιακά προγράμματα των κρατών μελών για την επόμενη περίοδο. Έχουμε τις γνωστές χώρες που έχουν υψηλό αριθμό συμβάντων Τι ε, ρόλο λοιπόν θα παίξει το ποσοστό σφάλματος για τα επιχειρησιακά προγράμματα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Εγώ λέω, Επίτροπε, να απαντήσετε στο τέλος σε όλες τις ερωτήσεις. Και τώρα θα πάρει το λόγο ο κύριος Ρούμπιχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια που αποφασίσαμε τον προπολογισμό του 2012 και 2013 νομίζω πως θα μπορέσουν να γίνουν όλες οι πληρωμές. Σημαντικό είναι να μας πείτε λοιπόν τι γίνεται με τις διαδικασίες αναστολής ε, πληρωμών. Πρακτικά από το 2009 για να δούμε πόσο αποτελεσματικά παρεμβαίνει το σύστημα. Κάποια νούμερα δηλαδή για να διαπιστώσουμε πως ε, η Κομισιόν κάνει τη δουλειά της βεβαίως. Μηδενικό ποσοστό σφάλματος σημαίνει μάλλον πως δεν γίνονται έλεγχοι, γιατί όταν γίνονται έλεγχοι ανακαλύπτουμε σφάλματα. Νομίζω λοιπόν πως ε, καλό είναι να δούμε σε βάθος χρόνου πώς έχει εξελιχθεί η κατάσταση με προειδοποιήσεις ε, και διορθώσεις και τι άποψη έχει το ελεγκτικό συνέδριο. Σας ευχαριστώ κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ε, να συγχαρώ τον κύριο Γκρέτεν για τον εκ νέου διορισμό του. Μετά, κύριε Επίτροπε, ε, πόσο καλά είναι τα, τα ελληνικά σας. Γιατί μας στείλατε τον κατάλογο των έργων στην Ελλάδα στα ελληνικά, για το οποίο σας ευχαριστώ. Αλλά ε, α, αν μπορείτε να μου το διαβάσετε, έτσι, γιατί αν δεν μπορείτε και εσείς να το διαβάσετε, δεν, δεν νομίζω ότι δεν μπορείτε να καταλάβετε τι γίνεται στην Ελλάδα, έτσι. Δεν φαντάζομαι να δουλεύει η Κομισιόν με αυτή τη λίστα έτσι, αλλιώς τουλάχιστον μία μετάφραση στα αγγλικά σε κάποια άλλη γλώσσα. Επίση. Οι απαντήσεις αυτές, το έγγραφο που μας στείλατε, πόσοι άνθρωποι τις έγραψαν. Εννοώ και από πόσες ε, γενικές διευθύνσεις ε, και τη... πρέπει να συμμετείχε νομίζω και κάποιες άλλες γενικές διευθύνσεις. Δεν είμαι ικανοποιημένη από τις απαντήσεις. Κάποιες ακούγονται ε, σατυρικές. Π.χ. η σελίδα 22 μας δίνεται α, απάντη... ρωτάμε έργα ποια έργα διαχειρίζεται συγκεκριμένα και η απάντηση είναι η Κομισιόν διαχειρίζεται προγράμματα και έργα. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Συχνά δηλαδή έχουμε την εμπειρία πως έχουμε πολύ στοχευμένες ερωτήσεις για το πώς λειτουργούν ε, τα πράγματα και μας, μας απαντάτε με γενικολογίες. Ε, η Κομισιόν διαχειρίζεται προγράμματα, Δεν ναι, το ξέρουμε αυτό, αλλά σας ρωτάμε συγκεκριμένα πράγματα. Το τέταρτο μου ερώτημα. τα, αυτό το οποίο περιγράψατε, επιστολές, προειδοποιητικές κτλ. Στο σελίδα 6 του ερωτηματολογίου αναφέρουμε, ε, βλέπουμε τον τίτλο ε, Παύσεις πληρωμών που ανακοινώθηκαν και εκεί πέρα είναι τελείως διαφορετικό το νούμερο από αυτό το οποίο μας αναφέρατε εσείς μετά. Έχουμε τους ε, φορείς ε, πιστοποίησης μετά μας λέτε πως ε, η Κομισιόν έχει λάβει 307, 304 από τις 317 αιτήσει εκθέσεις οποίες θα έπρεπε να έχει λάβει. 54 έλαβαν ε, άνευ ε, όρων διαβεβαίωση και οι υπόλοιπες είχαν ζητήματα. Οπότε Μιλάμε μόνο για ένα 46% το οποίο θεωρείται, στο οποίο θεωρείται πως υπάρχει η σωστή ε, παρακολούθηση. Θέλουμε λοιπόν πράγματι μια πιο στοχευμένη ε, προσέγγιση, αλλά εδώ πέρα αναφέρομαι στο ερώτημα Ε, στο οποίο που ανέφερα μετά, ε, ερώτημα 38, ε, 83, για την Ελλάδα, το οποίο αναφέρεται στην Task Force. Ε, οι απαντήσεις εδώ πέρα που δίνονται δεν έχουν ούτε μία σχέση με τις απαντήσεις που έδωσε η Task Force. Γιατί αυτό. Και μετά, ερώτηση 39. Μιλάμε για 1,13 ε, δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία ε, είχαν ε, παραμείνει από τον Απρίλιο του 2013 και δεν είχαν απορροφηθεί από την Ελλάδα. Τι έγιναν αυτά. Το ρωτήσαμε αυτό αλλά ούτε αυτή την απάντηση τη βλέπουμε σε αυτά τα οποία μας έδωσε η Κομισιόν. Και εδώ πέρα λοιπόν μια απάντηση μας οφείλεται. Thank you, Mr. Ευχαριστώ, Γκάιερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ σας ευχαριστώ για την δουλειά που κάνει το ελεγκτικό συνέδριο και εύχομαι καλή επιτυχία στα καθήκοντά σας στη νέα σας θητεία ένα ερώτημα προς το ελεγκτικό συνέδριο ο εισηγητής, ο κύριος Πίπερ, θέλει να έχει κάποιες εκθέσεις αναχώρα. Το αρέσει πάρα πολύ. Εγώ δεν ξέρω αν έχει κάποιο νόημα. Και ξέρω από την δικιά μου την εμπειρία ως συγητής πως το ελεγκτικό συνέδριο για διάφορους ε, λόγους ε, δεν είναι σε θέση να κάνει ε, μια γενική επισκόπηση για το ποσοστό σφάλματος. Κατά κανόνα κάνει κάποιες δειγματοληπτικούς ελέγχους και από εκεί πέρα εξάγει συμπεράσματα. Οπότε, αν είναι να δούμε το κατά πόσον έχει νόημα να κάνουμε εκθέσεις ένα χώρα, πρέπει να σκεφτούμε πως ε, εάν ταιριάζει καν με τον τρόπο λειτουργίας ε, του ελεγκτικού συνεδρίου. Δηλαδή πολύ απλά, σε πόσες χώρες κάνατε δειγματολοπτικούς ελέγχους στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής. Γιατί εντάξει γίνονται πολλά πράγματα με τα μαθηματικά, το αντιλαμβάνομαι, αλλά σε τελική ανάλυση το συνέδριο λέει πως ο πιθανό, το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος είναι 6,8, μπορεί να είναι λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, δεν μπορεί να αποκλείσει πως ε, το ποσοστό σε ένα κράτος μέλος που δεν έπεσε μέσα στο δείγμα μπορεί να είναι και ψηλότερο. Έτσι δεν μπορεί να το αποκλείσει. Οπότε, κύριε Γκρέτεν, εντάξει καταλαβαίνω τώρα πως είναι δύσκολο κι εσείς να απαντήσετε, αλλά κατά την άποψή σας πόσο χρήσιμες θα ήταν εκθέσεις αναχώρα δεδομένων και των περιορισμών που υπάρχουν στον τρόπο λειτουργίας του ελεγκτικού συνεδρίου γιατί οπωσδήποτε δεν νομίζω να μπορείτε να βάλετε κάτω από το μεγεθυντικό φακό όλες τις ε, χώρες. Και ε, αυτό βεβαίως ε, το ερώτημα απευθύνεται και προς την Κομισιόν. Όταν ήμουν και εγώ εισηγητής είδα το τι υπολογίζει το ελεγκτικό συνέδριο, το συνέκρινα με την Γενική Διεύθυνση περιφερειακής πολιτικής. Αν θυμάμαι καλά ήταν γύρω στα 18 κράτη-μέλη όπου ο ε, Γενικός Διευθυντής το προηγούμενο έτος λόγω ελήψεων στους ελέγχους ε, ήταν αναγκασμένος να πει πως αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να εγγυηθώ την κανονικότητα διεξαγωγής των προγραμμάτων. Έτσι 18 των τότε 27 ε, είναι πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Αν δει κανείς βεβαίως τις χώρες ε, μία προς μία ε, ήταν διαφορετικό το εύρος του φαινομένου, αλλά πριν περάσουμε σε μία απέτηση τέτοια ως κοινοβούλιο, εγώ θα ήθελα να γίνει μία συζήτηση. Για να μάθουμε δηλαδή ε, τι μπορούμε να έχουμε ως αποτελέσματα από αυτές τις ε, χώρες. Εντάξει, η παρομοίωση την οποία κάνατε με τον ΚΟΚ, εντάξει, καλή και έξυπνη, αλλά έχουμε τα μέσα από πλευράς ελεγκτικού συνεδρίου και κομισιών για να κάνουμε αυτά τα οποία θέλετε. Έχω τις αμφιβολίες μου. Και Εγώ θα έβαζα ένα ερωτηματικό, όπως σας είπα, στην απέτηση αυτή για εκθέσεις ε, αναχώρα. Τώρα, κύριε Ρούμπιχ, εγώ χαίρομαι για το ότι είχαμε αυτό το έγγραφο το οποίο ήταν εν μέρει αποτελεσμα και της δικής μου της ε, έκθεσης. Ε, βοήθησα και εγώ λιγάκι, αλλά θα ήθελα να πω το εξής. Χαίρομαι για το ότι θα έχουμε τις καθαρές διορθώσεις από το 2014. Ήταν κάτι το οποίο ζητούσα στην έκθεσή μου για την απαλλαγή. Τώρα θα προσπαθήσω λοιπόν να παγιδεύσω τον ε, Επίτροπο. Κύριε Χάν, έχετε κάποια αίσθηση του κατά πόσο θα μπορούσε να διορθωθεί εκ των υστέρων το ποσοστό σφάλματος μέσω των καθαρών αυτών διορθώσεων. Ε, ξέρω πως είναι δύσκολο να απαντήσετε, αλλά ισχυρίζεστε με σωστά επιχειρήματα πώς θα μπορούσε να είναι 0,8% το απευθύνεται προς το ελεγκτικό συνέδριο. Τώρα μιλήσατε για την διόρθωση την οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε εκ των υστέρων εάν είχαμε το, το μέσο. Ναι, είναι αποφασιστικό αυτό το νούμερο. Βλέπαμε κάποια ικανοποίηση πως η Κομισιόν δέχτηκε τις δικές μας τις απαιτήσεις για αναστελές πληρωμών με μεγάλη συνέπεια, αλλά πώς θα μπορέσουμε να προλάβουμε τα λάθη έτσι, δηλαδή η μείωση του ποσοστού σφάλματος, εντάξει, οφείλεται πραγματικά και στα νέα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Τα σφάλματα που έγιναν εντάξει οδήγησαν σε κάποιες ε, διακοπές Οι διακοπές χρηματοδότησης ε, βοηθάνε αλλά δεν ε, ρίχνουν το ποσοστό του σφάλματος Άρα θα πρέπει τα ελεγκτικά μέσα στο εθνικό επίπεδο να ενισχυθούν. Ε, εκεί πέρα υποστηρίζω πλήρως ε, τον εισηγητή. Δηλαδή όταν διαπιστώνουμε πως επιτόπου δεν εργάζονται επαρκώς οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, πρέπει να υπάρξει ένας αυτοματισμός. Να ε, διακόψει τις πληρωμές η Κομισιόν. Γνωρίζω βεβαίως πως τότε βρισκόμαστε σε ανταγωνισμό με τους πολιτικούς στόχους των κρατών μελών όταν δεν ρέει το χρήμα βεβαίως δεν εκπληρώνονται οι στόχοι τους οποίους έχουμε θέσει ως πολιτική, αλλά μετά Ω ελεγκτής του προπολογισμού λέω άμα είναι να πηγαίνουν στράφη καλύτερα να μην εκταμιεύονται τα λεφτά. Τελευταίο. ένα ερώτημα το οποίο σχετίζεται με την περσινή συζήτηση, κύριε Επίτροπε. Ο κύριος Γκρέτεν το υπογράμμισε. Οι κανόνες των ε, δημοσίων προμηθειών δεν είναι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι και εθνικοί κανόνες και παραβίαση των εθνικών κανόνων είναι ε, λάθος ε, βέβαια για το οποίο δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε την, ε, την Κομισιόν. Εντάξει τα γνωρίζουμε από την ε, Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία και το πώς φορτώνουν διάφορα πράγματα στο, στα έργα. Επίσης αν ξέρετε λοιπόν πόσο συνεισφέρει η παραβίαση των εθνικών κανόν στο ποσοστό τους, ε, του σφάλματος. Βεβαίως ε, θα θέλαμε και εδώ πέρα μια μελέτη, αλλά και αυτή η μελέτη θα είναι πάλι περιπτωσιολογία, γιατί κανείς δεν μπορεί να έχει γενική εικόνα της κατάστασης. Ίσως, δεν ξέρω, η Κομισιόν να έχει μια τέτοια εικόνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Σφόγγεν. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ζητήσω συγγνώμη γιατί κάθομαι κάπως σε χαμηλή καρέκλα. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω το ελεκτικό συνέδριο για την έκθεσή, της, έκθεσή του και την Επιτροπή. Έχετε μια βαριά ευθύνη γιατί τα χρήματα για την περιφερειακή πολιτική είναι από τα πλέον ορατά, τα πιο σημαντικά, τα πιο σημαντικά και γι' αυτό το λόγο ε, είναι σημαντικό και από την πλευρά μας η εκταμείευση των χρημάτων να γίνεται με σωστό τρόπο. Έχετε και εσείς με μεγάλη ευθύνη. εξετάσαμε, ε, μάλλον εξηγήσατε ποια είναι η αλλαγή στη μεθοδολογία και πώς θα γίνεται αυτή η καθαρή διόρθωση. Αλλά εδώ συζητάμε δύο διαφορετικά πράγματα. Το ελεκτικό συνέδριο χρησιμοποιεί κριτήρια Α και στις κριτήρια Β, διαφορετικά. Στόχος είναι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τους μεν και για τους δε. Νομίζω ότι ίσως θα ήταν πιο σκόπιμο να συζητήσουμε όλοι μαζί και να συμφωνήσουμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και του προπολογισμού. ορίζω επίσης το γεγονό ότι θα ότι μάλλον την προηγούμενη Παρασκευή δημοσιοποιήσατε την ανακοίνωσή σας για την καθαρή διόρθωση. Δεν πρόλαβα δημοσιονομική διόρθωση, δεν πρόλαβα να τη διαβάσω, θα το κάνω σύντομα. έχουμε συχνά την αίσθηση ότι αυτέ οι συζητήσει δεν είναι σημαντικέ επειδή αναφερόμαστε σε προηγούμενα οικονομικά αίτια, αλλά δεν ισχύει αυτό. Στην πραγματικότητα θα έπρεπε να αντλούμε διδάγματα από το παρελθόν και να τα εφαρμόσουμε αυτά τα διδάγματα στην επόμενη προγραμματική περίοδο, στα επόμενα χρόνια. Γιατί τα, τα ζητήματα που συζητάμε σήμερα είναι τα ίδια που είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν. Και πρέπει να δούμε κατά πόσον το σχέδιο δράσης για την περιφερειακή πολιτική βοήθησε και απλοποίησε τις διαδικασίες ε, ε, δημοσίων προημοφιών. Η απλοποίηση των διαδικασιών είναι κάτι που το συζητάμε κάθε χρόνο. Έχουμε διάφορες ιδέες για το πώς αυτή η απλοποίηση θα γίνει πραγματικότητα την επόμενη προγραμματική περίοδο. Τώρα έρχομαι σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Την ε, επόμενη προγραμματική περίοδο υπάρχουν και κάποιες προβλέψεις για την υποστήριξη των μικροπενσίων επιχειρήσεων αύξηση της, υποκρι... της ε, υποστήριξης αυτής. Όμως αυτή η αύξηση της υποστήριξης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορεί να ε, ε, νομοτελειακά μάλλον θα αυξήσει και τον αριθμό των οργανισμών που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα το ζήτημα της πρόβλεψης. Δεν μιλάμε πάντα για τους συνήθεις υπόπτους. Συχνά, για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει ανασταλεί η πληρωμή ε, των διαρθρωτικών ταμείων, όχι στην Ουαλία, όπως θα γνωρίζετε εκεί η κατάσταση είναι εξαιρετική, αλλά εξαιτία διοικητικών ε, ελήψεων έχουν ανασταλεί οι πληρωμές. Και ρωτώ πώς μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι όχι μόνο οι συνήθει αλλά και τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη θα έχουν στη διάθεσή του τι διοικητικέ υποδομέ που χρειάζονται για να αξιοποιούν τα διαρθρωτικά ταμεία και ε, να ε, ε, εκταμιεύονται και να χρησιμοποιούν τα χρήματα με τον σωστό τρόπο. Με ποιο τρόπο μπορούμε να το εξασφαλίσουμε αυτό. Ευχαριστώ κύριε Σόμπριχτ. Ευχαριστώ. Για άλλη μια φορά θα συζητήσουμε το ζήτημα τη απαλλαγή, αλλά τα ζητήματα είναι τα ίδια κάθε φορά. Και ήθελα να το επισημάνω αυτό, γιατί φαίνεται να μην μαθαίνουμε από το παρελθόν, από τα λάθη μας. Στο ζήτημα της απαλλαγής, το σημαντικό είναι ο τρόπος με τον οποίο κατανεμήθηκαν οι πόροι ή η αποτελεσματικότητα. Κατά την άποψή μου, είναι Πρώτα απ' όλα σημαντικό να συζητάμε για την αποτελεσματικότητα και μετά για την ορθή κατανομή των πιστώσεων. Γιατί συχνά μπορεί να γίνονται οι ε, χρηματοδοτήσεις με τρόπο ε, νομότυπο αλλά να μην είναι αποτελεσματικές. Η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου εξελίσσεται κατά τη διάρκεια των ετών, μας δίνει νέες πληροφορίες, αλλά τα προβλήματα που αναδεικνύει παραμένουν τα ίδια. Βεβαίως και εκτιμώ την, ε, το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη συνεργασία της με, τον, με το λεκτικό συνέδριο, αλλά το ερώτημα είναι ποιον ελέγχουμε τελικά. Ελέγχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ελέγχουμε τα κράτη-μέλη ή το κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήλεγξε σωστά τα κράτη-μέλη. Το ίδιο ερώτημα έχουμε εδώ και χρόνια. Και πρέπει κάποια στιγμή να το απαντήσουμε με τρόπο σαφή. Όταν το ελεκτικό συνέδριο κάνει ένα δειγματοληπτικό έλεγχο και προτείνει δημοσιονομικές διορθώσεις, αυτές δεν είναι τιμωρητικού χαρακτήρα, πρόκειται για δημοσιονομικές διορθώσεις. Στο τέλος του έτους πρέπει να ελέγχουμε ε, και να σχηματίζουμε τη συνολική εικόνα ή μήπως θα ήταν καλύτερα αυτός ο έλεγχος να γίνεται αμέσως από τη στιγμή που διαπιστώνεται μια ε, παρατυπία. Με άλλα λόγια, προσπαθούμε να αξιολογήσουμε συνολικά την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας αυτού του μηχανισμού ή απλώς λαμβάνουμε μια φωτογραφία σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Είμαι σιώδης εισηγητής για την απαλλαγή ε, εκ μέρους της Επιτροπής ε, Περιφερειακής Πολιτικής. Κάθε έτος εκφράζουμε την πολιτική μας άποψη για τους μακροπρόθεσμους στόχους και ζητούμε αλλαγές. Αυτό οδηγεί στο να λέμε κάθε χρόνο ότι υπήρξαν κάποιες βελτιώσεις, η κατάσταση ε, έχει βελτιωθεί αλλά παραμένουν λάθη, παραμένουν προβλήματα. Οι βελτιώσεις αυτές έχουν προεκύψει από το σχέδιο δράσης. και πιστεύω ότι η νομοθεσία έχει οδηγήσει σε αυτές τις βελτιώσεις. Με άλλα λόγια, πιστεύω ότι έχει σημειωθεί πρόοδο παρά το γεγονό ότι παραμένουν κάποιες παρατυπίες. Αλλά εγώ θέλω να θέσω δύο ερωτήματα στον Επίτροπο. Εξηγήστε μου το εξή. Είπατε στο λόγο σας Ζητώ συγγνώμη που δεν άκουσα όλη την παρέμβαση του εισηγητή γιατί άργησα, αλλά πάντως άκουσα όλη την παρέμβαση του Επιτρόπου. Είπατε λοιπόν ότι υπάρχουν δημοσιονομικέ διορθώσει και από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την πλευρά του Συμβουλίου. Θέλω όμω να μου δώσετε περισσότερε λεπτομέρειε. Ποια είναι η θέση της Επιτροπής για τις καταποκοπήν δημοσιονομικές διορθώσεις. Και τώρα έρχομαι στο μέλλον, όχι για την απαλλαγή την τρέχουσα, αλλά στο μέλλον. Έχετε προτείνει καινοτόμε δράσεις στο πλαίσιο τη περιφερειακή πολιτική. Δεν μιλάω για τις δράσεις για την καινοτομία, μιλάω για τις καινοτόμε δράσει. Innovative action, όπω τα λέτε στα αγγλικά, για τι ε, αστικέ περιοχέ. Καινοτομία σημαίνει κίνδυνος, σημαίνει αφεβαιότητα, σημαίνει ότι εκφεύγουμε τα συνηθισμένα. Άρα, κύριε Επίτροπε, θεωρείτε μήπως ότι θα πρέπει να αλλάξουμε και εμείς την προσέγγιση μας όσον αφορά τον έλεγχο της ε, χρήσης των πόρων για αυτές τις καινοτόμες δράσεις. Μήπως θα θέλατε να αυξηθεί το επιτρεπόμενο περιθώριο ασφάλματος για εκείνες τις καινοτόμες δράσεις. Ευχαριστώ κύριο Σόντερκα. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και εγώ το ελεκτικό συνέδριο και τον Επίτροπο Χάν για όλες τις διευκρινήσεις που μας έδωσε. Επίσης και για αυτά που είπατε για, τα... για το Ταμείο Αλληλεγγύης. Ωστόσο, ορισμένε από τι απαντήσει σα εγείρουν νέα ερωτήματα. Και άλλε, στην πραγματικότητα φωτίζουν τον λόγο για τον οποίο υπήρχαν κάποια από τα προβλήματα που είχαμε στο παρελθόν. Καλό θα ήταν να τα είχαμε αυτά τα στοιχεία πιο νωρί, αλλά εν πάση περιπτώσει καλώ τα αποκτήσαμε τώρα. Σε δύο θέματα θα σταθώ εγώ σήμερα. την ε, κακή χρήση των πόρων του Ταμείου Αλληλεγγύης και την παραβίαση της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις. Ας συζητήσουμε πρώτα απ' όλα για το ζήτημα των ατασταλιών ε, ευρωπαϊκών πόρων. Αυτό δεν είναι ένα ζήτημα μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπή, είναι ένα ζήτημα μεταξύ ε, Ελεκτικού Συνεδρίου και Επιτροπή. Συμφωνώ πλήρω με το Ελεκτικό Συνέδριο όταν λένε ότι το ε, Ταμείο Ελληνικής έχει εξαιρετικά και μεγάλη σημασία. Μιλάμε για 60 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για έργα που αφορούσαν κυρίως λίγους και όχι ε, για περισσότερα έργα που θα αφορούσαν περισσότερους πολίτες. Το τομέα της στέγασης. Και να το να δημιουργηθούν γούνται ε, ε, οι οποίες να έχουν κακές συνθήκες στην πραγματικότητα δυσχεραίνει την κατάσταση, δεν είναι βελτίωση. Και το δέχτηκε αυτό η Επιτροπή δεχόμενη ότι με χρήση των πόρων των Ταμείων Αλληλεγγύης θα χτίζονται λιγότερες εστίες ε, με α, καλύτερες συνθήκες θα μπορούσαν μάλιστα να είχαν δώσει τη χρηματοδότηση ε, σε ακόμα περισσότερες αν είχαν δεχθεί ε, προσωρινές, ε, προσωρινά κτίσματα. Το ερώτημα είναι τι είναι προσωρινό. 30, 40, 60 χρόνια. χωρίς ανοικοδόμηση. Δεν μονιμότερο του προσωρινού. Επομένω, θα ήθελα να μου εξηγήσετε λίγο καλύτερα με ποια έννοια ε, ε, αντιλαμβάνεται την προσωρινή στέγαση η Επιτροπή. Επίσης θα Ήθελα η Επιτροπή να μου εξηγήσει πώς προκύπτει αυτή η διαφορά. Και αν δεν μπορεί να μας την εξηγήσει η Επιτροπή, μήπως καλύτερα να προσφύγουμε στο ελεκτικό συνέδριο. Η θέση του ελεκτικού συνεδρίου ήταν πιο σαφής. Ένα άλλο ζήτημα είναι το γεγονός ότι η οδηγία υπερηδημοσίων συμβάσεων δεν έχει πλήρω εφαρμοστεί η μεταγραφή πλήρω στα κράτη-μέλη. Και φαίνεται ότι η Επιτροπή έχει αποφύγει να αγγίξει το ζήτημα της ανοικοδόμησης σπιτιών μετά από σεισμούς. Η ανοικοδόμηση λοιπόν και οι απαλατριώσεις αφορούσαν ποσό περίπου 920 εκατομμύρια ευρώ. Και τα 450 προέλθαν από το Ταμείο Αλληλεγγύης, το υπόλοιπο από την Ιταλία. Τώρα πέρα από αυτή τη χρήση των 920 εκατομμύριων ευρώ, πέρα από αυτές, η Επιτροπή είπε ότι διαπίστωσε ατασταλίες όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις τουλάχιστον 306 εκατομμύρια ευρώ. Το 1 τρίτο δηλαδή του συνολικού ποσού. Ατασταλίες λοιπόν σε τεράστιο βαθμό που δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να τύχουν έγκριση ε, με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Μιλάμε για το 1 τρίτο το 60% του ποσού που είχε προβλέψει ως πίστοση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάθε φορά που διαπιστωνόταν μια παρατυπία, αυτό το ποσό το εγγράφαμε υπό το ποσό που προερχόταν από την Ιταλία. πάνω από 70% ε, καταλήγουμε τελικά. Και αυτό δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να γίνει δεκτό με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και η Επιτροπή μας λέει ότι εδώ δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά το ερώτημα που θέτω εγώ είναι λογικό αυτό. Είναι ότι τρόπος με τον οποίο θα έπρεπε να πορευόμαστε. Και το θέτω αυτό. Γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ομάδες οργανωμένου εγκλήματος οι οποίες αξιοποιούν τα παραθυράκια στον νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις για τους δικούς τους σκοπούς. Ε, φυσικά Γνωρίζω ότι δεν πρόκειται όλες οι όλα τα λάθη δεν είναι ατασταλείς και δεν είναι όλες οι ατασταλείς εγκλήματα. Τα γνωρίζω αυτά. Και είναι εξαιρετικά προσεκτικές οι διατυπώσεις ε, και του ελεκτικού ε, συνεδρίου και της Επιτροπής. Αλλά υπάρχει τεράστιος κίνδυνος απάτης. Ένα άλλο πρόβλημα που παραμένει με όλα αυτά είναι ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιο ποσοστό των ευρωπαϊκών πόρων τελικά ε, δόθη για τους σκοπούς που είχαν προβλεφθεί. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τελικά ποια ήταν η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε να έχουμε μια αίσθηση ότι η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν, ήταν τεράστια, αλλά τελικά δεν μπορούμε να την ποσοτικοποιήσουμε. Και εν πάση περιπτώσει το θεωρώ απαράδεκτο απλώ να μεταβιβάζουμε τις, τα ποσά των λαθών από το ένα κονδύλιο στο άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή για, την, για τις εξηγήσει. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι από τον κύριο Γκρέτεν. Το ελεγκτικό συνέδριο θα ήθελα να μου πει ποιος είναι, ποιο είναι το συγκεκριμένο ποσοστό έλλειψη σεβασμού με τους κανόνες. Μιλάμε για τις σοβαρές παρατυπίες. Και επιπλέον, με βάση ποια κριτήρια χαρακτηρίζεται σοβαρές τις παρατυπίες. Και επιπλέον, τα λάθη αυτά, οι σοβαρές αυτές παρατυπίες, οι σοβαρές μη συμμορφώσεις, οφείλονται στα κράτη-μέλη ή στην Κομισιόν περισσότερο. Επίση, σε ό,τι αφορά τι διορθώσει και τι αναστολέ. φέτος βλέπω ότι υπάρχει μια υποσημείωση με νούμερα. Ε, στην πραγματικότητα διαβάζουμε το κείμενο, δεν καταλαβαίνουμε και να διαβάσουμε τι λεπτομέρειε τις λεπτομέρειες για να καταλάβουμε τι τρέχει. Οι οικονομικές διορθώσεις για το 2012. Στα πλαίσια της κοινή ε, διαχείρισης υπάρχει ένα νούμερο για την Ισπανία. Για την ε, Ισπανία νομίζω ότι τα πράγματα είναι τραγικά. Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι οι εξηγήσει που μας δώσατε. Αυτές οι διορθώσεις έγιναν πριν από το 2010 υποτίθεται. Αλλά τώρα το... βλέπω ότι τα νούμερα είναι ακόμα... των λαθών ας πούμε είναι ακόμα μεγαλύτερα. Αυτά που συμβαίνουν στην Ισπανία είναι τραγικά. Όταν βλέπουμε τις διορθώσεις όμως ε, βλέπουμε ότι εντάξει πρέπει να σχετικοποιήσουμε τα πράγματα. Χρειάζομαι και άλλες εξηγήσεις γιατί αλλιώς δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Αν πάρουμε την ίδια περίοδο, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010 είχαμε 104 περιπτώσεις ανοιχτές στην Γερμανία, λιγότερες στην Ισπανία, αλλά τώρα εμείς έχουμε ξεπεράσει τη Γερμανία. Μας εξηγείτε παρακαλώ πώς φτάσατε σε αυτούς τους υπολογισμού. Επίσης βλέπω τα διάφορα προγράμματα. Γερμανία, προγράμματα που αναστάλησαν Ταμείο ε, Συνοχής και ΦΕΝΤΕΡ. 31 Δεκεμβρίου 2012. Έχουμε δύο γερμανικά προγράμματα, μάλλον διορθώνει η μιλήτρια, ένα γερμανικό και ένα ιταλικό που έχουμε ανασταλεί. Τελικά, ε, έχει ανασταλεί προσωρινά ή απλώς το παραπέμψαμε σκαλένδες αυτό το γερμανικό πρόγραμμα. Θα θέλαμε το συνέδριο να μας δίνει εκθέσεις αναχώρα και να βάζει βαθμολογίες, κακές και καλές στις χώρες. Εδώ μιλάμε για περιφερειοποίηση, ε, για διακυβερνητικό επίπεδο διαχείρισης. Υπάρχει πουθενά η το κοινοτικό πνεύμα. αν έχουμε μία έκθεση αναχώρα, και αν ο στόχος είναι η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ όλων, τότε πραγματικά δεν βλέπω πώς θα τα καταφέρουμε. Μιλάμε για ευρωπαϊκά προγράμματα, μιλάμε για εθνικά προγράμματα. Όχι, μιλάμε για εθνικά προγράμματα. Έχουμε το Interreg, έχουμε διάφορα προγράμματα. Αυτά πώς μπορούμε να τα δούμε. Μπορούμε να τα θεωρήσουμε, ας πούμε, πολυετή ευρωπαϊκά προγράμματα. Μία τελική ερώτηση έχω εγώ. Βλέπω μια διαφορετική άποψη μεταξύ συνεδρίου και κομισιών για τα ε, σφάλματα. Το συνέδριο λέει ότι αν γίνει διόρθωση από τη Κομισιόν μέσα στην ε, χρονιά, αυτό το λάθος δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ενώ η Κομισιόν θεωρεί αντίθετα ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτή η διόρθωση. Προφανώς. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε λοιπόν αυτό το, ακόμα μια φορά το σημείο. Κομισιόν. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι δεν μπορείτε να παραπονεθείτε ότι δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο αυτά που λέτε. Αυτό το θέμα προκαλεί τρομερό ενδιαφέρον. Προφανώς, αλλά το περίμενα κιόλας, ε, μην νομίζετε. Ναι. Θα προσπαθήσω να απαντήσω με τη σειρά, αλλά υπάρχουν πολλά ερωτήματα που επαναλαμβάνονται. Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Πίπερ για αυτοματισμό. Προσπαθούμε να τυποποιήσουμε για διάφορους λόγους. Αλλά βεβαίως πάντα υπάρχει κάποιο περιθώριο. Αλλά μπορώ να σας πω πως όταν ένα κράτος μέλος ε, έχει σε εθνικές ε, ελληνικές αρχές ε, ποσοστό σφάλματος πάνω από 2% κινητοποιούμαστε. και μετά αναλόγως προχωράμε σε διακοπές και αναστολές. Και κύρια Γελασέντερ, ναι, κα, είναι πράγματι προσωρινά αυτά. Αυτός είναι ο στόχος. Αλλά εάν μέχρι το τέλος της περίοδου δεν έχει λυθεί το ζήτημα, υπάρχουν και καθαρές διορθώσεις. Αλλά σκοπός μας είναι να είναι προσωρινά αυτά τα μέτρα. Για να επανέλθω στον κύριο Πίπερ, έχουμε 15 κράτη-μέλη όπου ε, ξέρουμε με βάση την αξιολόγηση κινδύνου πως πρέπει να δούμε πως έχει απόδοση και στον τομέα του ελέγχου. Και Αυτό είναι κάτι βεβαίως το οποίο μπορεί να αλλάξει. Αν μετά από μερικά χρόνια έχουμε τη βεβαιότητα πως οι δομές ε, λειτουργούν, τότε βεβαίως ε, αποσυρώμαστε έτσι. Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε και τους ανθρώπινους πόρους που έχουμε αποτελεσματικά. Από 700 υπαλλήλους στη Γενική Διεύθυνση Ήδη έχουμε 83 που ασχολούνται αποκλειστικά με τον έλεγχο. Ε, γύρω στο 12% του προσωπικού. Έχουμε φτάσει λοιπόν ένα κάποιο επίπεδο που έχουμε μια ισορροπία μεταξύ ελέγχου και παραγωγής, απόδοσης θα έλεγα και νομίζω πως ε, έχουμε συνολικά 2.600 ε, ισοδύναμους ε, πλήρους απασχόλησης ε, θα έλεγα στον τομέα αυτόν οπότε προσπαθούμε όπως είπα να βρούμε αυτή την ισορροπία γι' αυτό το οποίο πρότεινε ο κύριος Ρούμπιχ νομίζω μπορούμε να σας δώσουμε έναν κατάλογο διακοπών και αναστολών αναχώρα Τώρα, η κυρία Γκρέσλε Εντάξει, καταλαβαίνω, σας στείλαμε κάτι στα ελληνικά. Συγγνώμη. Αλλά απ' την άλλη, να σας πω, ε, ειλικρινώς προσπαθήσαμε να απαντήσουμε πάρα πολύ γρήγορα και πράγματι οι αρμόδιοι για την Ελλάδα βεβαίω ξέρουν ελληνικά, Έλληνες ή Κύπροι. Έτσι. Και επειδή η επικοινωνία για αυτά τα ζητήματα ε, γίνεται στα ελληνικά και επειδή μάλλον εσείς λάβατε τις πληροφορίες αυτές από δεύτερο χέρι, για λόγους ταχύτητας δεν καταφέραμε να έχουμε μια επίσημη μετάφραση. Ε, υποθέτω πως ε, μπορεί κάποιος ε, από το κόμμα σας ε, να σας τα εξηγήσει. Αλλά τέλος πάντων θα προσπαθήσουμε στο μέλλον να σας τα... θα σας τα στείλουμε δηλαδή στο μέλλον, αλλά υποθέτω πως έγινε κάποιο λάθος λόγω διασύνης. Μας περιπτώσει είναι μια επίσημη γλώσσα με την οποία επικοινωνούμε με τα κράτη-μέλη, έτσι. Όσον αφορά τώρα τα διάφορα νούμερα. Δεν μπόρεσα να τα παρακολουθήσω. Υποθέτω πως εάν δει κανείς τα χρόνια, νομίζω πρέπει να ταιριάζουν τα νούμερα, αλλά θα τα επαληθεύσω. Ε, υπάρχει όμως συχνά μια... διαφορά εάν θέλετε μεταξύ των ε, δειγματοληπτικών στοιχείων και των ε, στοιχείων που δίνουμε στις απαντήσεις μας, τα οποία είναι πάντα τα πιο πρόσφατα και τα πιο επίκαιρα. Δεν ξέρω ίσως να οφείλεται και στο, σε ποιο χρονικό σημείο έγιναν διαθέσιμα τα πιο ε, τελευταία στοιχεία. Αλλά υπάρχουν ε, πράγματι και σε διαφορετικές επιτροπές σε διαφορετικά στοιχεία ανάλογα με το πότε έγινε η ερώτηση και πότε απαντήθηκε πράγματι. Για το 38 και 39 θα το δούμε γραπτός και θα το διευκρινίσουμε οπωσδήποτε. Κύριε Γκάιερ για τις καθαρές διορθώσεις. Σας ευχαριστώ και για αυτό το οποίο μου είπατε αλλά κοιτάξτε, τι μπορούμε να πούμε γύρω στα δύο τρίτα των ε, σφαλμάτων ε, τα ανακαλύπτουν οι εθνικές ελεγκτικές αρχές. Δηλαδή επί της αρχής πράγματι λειτουργούν καλά και σε γενικές γραμμές θα ήθελα να το πω και εδώ πέρα πως Έχουμε σε γενικές γραμμές μεγάλη εμπιστοσύνη στην επαγγελματική επάρκεια των ελεκτικών αρχών στα κράτη-μέλη. Εκεί όπου έχουμε ανησυχίες είναι είτε για την επαρκή στελέχωση, αναφέρθηκε το είπατε και εσείς για την Αγγλία, υπάρχουν και άλλα παραδείγματα, ή για την επαρκή ανεξαρτησία. Αυτές είναι οι βασικές μας ανησυχίες ε, που πρέπει να δούμε είναι λοιπόν ζητήματα τα οποία στο μέλλον θα μπουν όσον αφορά την αιρεσιμότητα την εξάντε. Αλλά αν δούμε ήδη πως δύο τρίτα ανακαλύπτουν, τα ανακαλύπτουν οι εθνικές αρχές και το ένα τρίτο το ελεγκτικό συνέδριο ή εμείς, ε, πράγματι υπάρχει δυνατότητα βελτιώσεων ε, εάν μέσω του αποτρεπτικού χαρακτήρα των καθαρών ε, διορθώσεων γίνουν πιο προσεκτικές οι εθνικές ελεγκτικές αρχές. Τώρα το τι επίδραση θα έχει ακριβώς το ποσοστό σφάλματος δεν μπορώ να σας το πω αλλά νομίζω υπάρχει, υπάρχουν αρκετές δυνατότητες. Τώρα, για τις δημόσιες προμήθειες, ε, νομίζω ο κύριος Μπαρνιέ θα υποβάλει μία πρόταση για νέες κατευθυντήρες γραμμές, οι οποίες θα οδηγήσουν σε απλοποίηση των πραγμάτων, έτσι ώστε να μειωθούν, νομίζω, ή να μειωθούν τα ποσοστά ασφαλμάτων. Πράγματι, να απαντήσω και στον κύριο Φων, είναι αυτή μια πρόκληση για το μέλλον. Δηλαδή, αν θέλουμε να διαθέσουμε διπλά μέσα, διπλάσια μέσα από ό,τι τώρα για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οπωσδήποτε θα αυξηθούν οι το ύψος της κάθε μίας ενίσχυσης ε, και βεβαίως η δουλειά των διαχειριστικών αρχών και προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό με απλοποιημένες διαδικασίες με περαιτέρω απλοποίηση υπομορφήν ε, διευρυμένων ε, δυνατοτήτων ε, καταποκοπήν υπολογισμών αλλά πρέπει βεβαίως να παραδεχτούμε πως είναι μια νέα πρόκληση ε, θα είναι μια νέα πρόκληση για το πρώτο επίπεδο αυξημένος αυτός αριθμός ε, έργων. Αλλά αυτό είναι αντικείμενο της ε, εξάντε Ο κ. Σόλμπριχτ αναφέρθηκε στις διαβουλεύσεις εντός της Επιτροπής σας. Εγώ θεωρώ και είμαι πεπισμένος πως ειδικά όσον αφορά την, ε, το σχέδιο δράσης της Επιτροπής σας ε, είχαμε δραστικές ε, βελτιώσεις της απόδοσης de facto νομίζω είχαμε μία μείωση στο μισό του ποσοστού σφάλματος και αν δούμε τον όγκο των πληρωμών, το ότι αυξάνονται τα έργα και ταυτόχρονα το επίπεδο των ε, σφαλμάτων ε, μειώνεται, νομίζω δείχνει πως ε, υπάρχει μία τάση χρόνο το χρόνο να εξελισσόμαστε εμείς και τα, και τα κράτη-μέλη έτσι. Οπότε βλέπω εγώ συνολικά μια θετική τάση. Και βεβαίως ε, θα χαιρόμουν να αναφερθεί και στα συμπεράσματα. Τον ε, κύριο Σόντρικαρτ πράγματι αυτό το οποίο είπατε είναι κάτι το οποίο υπάρχει όντως ε, στην απαλλαγή Για το Αμπρούτσο το θέμα που αναφέρεται οπωσδήποτε προσωρινό δεν είναι 50-60 χρόνια έτσι. Αλλά από πλευράς ε, όγκου ε, ε, εντάξει και δεδομένου των τοπικών ε, ιδιαιτεροτήτων υπάρχει κάποια ευελιξία. Εντάξει βεβαίως μιλάμε για ένα λογικό διάστημα 5 ετών ε, σε αυτή την ιδιαίτερη κατάσταση όπου είχαμε χιλιάδες αστέγους και έπρεπε άμεσα να έχουν ε, προσωρινό κατάλημα. Ε, εντάξει, όταν έχουμε τέτοιες ε, καταστάσεις ανάγκης όπου πρώτα απ' όλα προέχει η προστασία των ανθρώπων Εντάξει, μπορεί να μην έγιναν όλα μέχρι κεραία ε, σύμφωνα με τον κανονισμό, αλλά εκεί πέρα πραγματικά ζητάω την κατανόησή σας. Και αυτό δεν βεβαίως δεν αλλάζει σε τίποτα το ότι στον έλεγχο θα τα δούμε όλα μέχρι κεραία. Γι' αυτό ακριβώς είχαμε 300 εκατομμύρια ευρώ τα οποία δεν δεχτήκαμε να πληρώσουμε και ε, στο πλαίσιο του εφικτού κινείται αυτό, έτσι, γιατί αυτό είναι ένα πολύ μικρότερο κομμάτι των συνολικών πληρωμών που διατέθηκαν από την Ιταλική πλευρά, έτσι, κατά κύριο λόγο. Οπότε και με την αφαίρεση αυτή νομίζω των 5 ε, εκατομμυρίων ε, είχαμε 305 εκατομμυρίων είχαμε ε, πολύ περισσότερα ε, λεφτά τα οποία εισέρευσαν. Οπότε εντάξει μπορεί να διαφωνούμε σε αρκετά πράγματα αλλά νομίζω πως ε, τώρα να υποψιάζεστε τους συνεργάτες μου πως συνεργάζονται με τη μαφία κάπου παραπάει. Δεν ξέρω αν σας κατάλαβα και σωστά, έτσι. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, πως οι συνεργάτες μου εργάζονται και έχουν καθαρή την ε, συνείδησή τους, δεν ε, εργάζονται και στο 8ωρο, φεύγουν ειδικά όσον αφορά το Ταμείο Αλληλεγγύης, έτσι. Ήθελα να, το πω αυτό εδώ πέρα. Και κυρία Γιάλα Σέντερ την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε μια παρουσίαση για την ακριβή περιγραφή του όρου ε, σοβαρές ελλείψεις στο πλαίσιο ακριβώς των πράξεων κατ' έτσι ώστε πράγματι να υπάρχει σαφήνεια Έχετε δίκιο πράγματι στο παρελθόν, στο Interreg είναι κάπως δύσκολα τα πράγματα και δεν μπορούν να γίνουν εκθέσεις ανά χώρα. Υπάρχει μια συνολική έκθεση για το Interreg και πρέπει πράγματι να το δούμε αυτό το ζήτημα. Συνοψίζοντας λοιπόν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την θετική κριτική σας. Και για να επανέλθω σε κάτι που ρώτησε ο κύριος Πίπερ στην αρχή. Οπωσδήποτε ε, όταν κάποιος βεβαίως παραβιάζει συνέχεια τους κανόνες ε, θα έχει μετά στο τέλος υψηλότερη δημοσιονομική διόρθωση. Δηλαδή μιλάμε για έναν διπλασιασμό όταν πρόκειται για υπότροπους. Αλλά οι λεπτομέρειες ε, θα φανούν ε, στην πράξη κατεξιοδότηση. Και μια τελευταία παρατήρηση. Μπορεί εάν δει κανείς μόνο τις χώρες, γιατί υπάρχουν χώρες όπου υπάρχει η εντύπωση πως είναι η συνήθις ύποπτη. Αλλά εάν μπει στην ουσία και στις λεπτομέρειες, διαπιστώνει πως ε, στις χώρες από χρόνο σε χρόνο υπάρχουν διαφορετικές ε, διαχειριστικές αρχές που είναι υπεύθυνε για το ποσοστό του σφάλματος, όπως παραδείγματο χάρη η Ισπανία. Η Ισπανία πράγματι έχει πολύ πολύπλοκη δομή. Εδώ πέρα νομίζω θα συμφωνήσετε. Και ελπίζω στην επόμενη περίοδο μαζί με την Ισπανική κυβέρνηση και τις περιφέρειες να υπάρξει κάποια απλοποίηση. Γιατί και αυτό είναι ποινή, ε, πηγή με των ε, συνεχών λαθών. Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικές ε, διαχειριστικές αρχές ε, πλην εξαιρέσεων που ε, δημιουργούν τα νέα λάθη και οι ελεγκτικές αρχές είναι αυτές οι οποίες τελικά είναι αξιόπιστες και πάνω σε αυτές νομίζω μπορούμε να βασιστούμε. Σας ευχαριστώ. Το ελεγκτικό συνέδριο, μήπως θα ήθελα να προσθέσει κάτι. Σύντομα παρακαλώ όμως. Δύσκολο πρόεδρε. Υπήρξαν ερωτήσεις για τις ε, οικονομικές διορθώσεις και ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ του συνεδρίου και της Επιτροπής. Όπως είπα και πριν, το συνέδριο είναι υποχρεωμένο στην ετήσια έκθεση να μιλήσει για το αν οι συναλλαγές είναι νόμιμες και κανονικές. Η Κομισιόν προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η προσέγγιση των δύο είναι διαφορετική, αλλά συμπληρωματική όμως. Το συνέδριο λαμβάνει υπόψη τις δημοσιονομικές διορθώσεις και τις ανακτήσεις και τις λεπτομερείς διορθώσεις σε επίπεδο έργο. Δηλαδή, ε, τμήμα του έργου ή έργα τα οποία ε, δεν συμμετέχουν στην τελική έκθεση, ας πούμε. Όταν δεν έχουμε τα ακριβές ποσό των παράτυπων δαπανών στις δηλώσεις, ε, εκεί δεν ε, αυτή, αυτό το λάθος δεν επηρεάζει το συνολικό ποσοστό του λάθους. Το κράτος μέλος είναι υπεύθυνο να μιλήσει για αυτά τα θέματα και να διορθώσει ε, αυτά τα προβλήματα. Ε, το κράτος μέλος, αν δηλαδή η δημοσιονομική διόρθωση θα αφορά το ίδιο το έργο. Αν το κράτος μέλος δεν κάνει τη δημοσιονομική διόρθωση επίπεδο έργου, τότε ένα τμήμα της κοινή διαχείρισης δεν έχει γίνει και το συνέδριο δεν μπορεί να αποδείξει ότι αυτές οι διορθώσεις επηρεάζουν τα επίπεδα λαθών στις ε, συναλλαγές. Αυτή είναι η προσέγγισή μας στις ε, δημοσιονομικές διορθώσεις και αυτό εξηγεί το γιατί έχουμε διαφορές με την ε, Κομισιόν. Αυτό για το ερώτημα αυτό που μου θέσατε για τις δημοσιονομικές διορθώσεις ήθελε βεβαίως ε, να με φέρει σε δύσκολη θέση, κάτι το οποίο δεν είναι βεβαίως ε, και κίνδυνο. Κοιτάξτε, θα ήθελα εγώ να πω πως σε 17 κράτη-μέλη ε, τα οποία εξετάσαμε, θα τα βρείτε αυτά στην παράγραφο 5, 25, και είναι νομίζω και, κοιτάξτε δεν είναι αντιπροσωπευτικό για όλα τα κράτη-μέλη. Εμείς λειτουργούμε στατιστικά. Εάν εξετάζαμε το Λουξεμβούργο θα έπρεπε να εξετάσουμε 180 προγράμματα. Δεν υπάρχουν 180 προγράμματα στο Λουξεμβούργο ή στη Μάλτα. Έτσι θα έπρεπε να εξετάσουμε όλα τα έργα. Μιλάμε για έργο συσήφιο. Έχουμε 900 ε, υπαλλήλους, θα χρειαζόμασταν ε, άλλους 1800. Ε, δεν έχει νόημα, έτσι. Αλλά υπάρχουν μόνο τέσσερις χώρες που κάνουν αυτές τις, τις εκθέσεις. Αυτό το 2013 ήταν Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, Σουηδία και Δανία είδαμε τις εκθέσεις δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του ελεγκτικού συνεδρίου, αλλά εξετάζουμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για την δουλειά μας. Και θα, θα τοποθετηθούμε. Η κυρία Γιάλα Σέντερ ρώτησε για το ποσοστό σφάλματος. Έχουμε 31% όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες, 31% ε, παραβιάσεις, διαπιστώσει, 12% σοβαρές, δηλαδή παραβιάσεις όπου, παραδείγματος χάρη, ε, είχε περιοριστεί η διαδικασία του διαγωνισμού, δεν ήταν ανοιχτός ο διαγωνισμός, δεν ήταν ε, η διακήρυξη πανευρωπαϊκή. Τα βλέπετε αυτά στο κουτί 5.1 της έκθεσής μας. Επίσης για εμάς σοβαρή παραβίαση είναι όταν το αποτέλεσμα της ε, προκήρυξης ε, θα έπρεπε να είναι διαφορετικό. Και όταν διαπιστώνουμε Ε, λιγότερο σοβαρέ ε, παραβιάσεις είναι ε, τελείως διαδικαστικά τα ζητήματα και αυτό είναι στην παράγραφο 534. Αυτά εν ολίγη κύριε Πρόεδρε, αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις ευχαριστώ να απαντήσω γραπτό. Ευχαριστώ. Κυρία Κρέσλερ. Με συγχωρείτε κύριε Επίτροπε, αλλά έχω πρόβλημα αρχή. Δηλαδή αν είναι να επιτύχουμε τους πολιτικούς μας στόχους, να μην έχουμε κανέναν ε, έλεγχο και θα είναι όλα υπέροχα. Αλλά εγώ δεν έχω εντύπωση πως θα επιτύχουμε τους πολιτικούς στόχους. Θα ήθελα να υπενθυμίσω πως οι αιτήσεις εκθέσεις έλεγχου είναι ε, σημαντικές, αλλά τι μπορούμε να πούμε όταν από τις... 317 ε, ε, εκθέσεις, γύρω στις μισές 114 μόνο έχουν ελεγχθεί. Επίσης όταν μιλάτε για 2.600 ε, άτομα τα οποία θα παίρνουν ετήσιο μισθό 50.000 ε, έχουμε ένα 3-4% κόστος ε, του ελέγχου. Οπότε αυτό το οποίο λέτε ότι κοστίζει πάρα πολύ δεν με πείθει. Κύριε Επίτροπε, όχι, εγώ δεν είπα ότι κοστίζει πάρα πολύ, απλά ε, μίλησα για μια συγκεκριμένη ισορροπία μεταξύ ελέγχου και ε, τελικά αποτελέσματος, έτσι. Δηλαδή, όπου και αν πηγαίνω, ε, εντάξει, δεν με βασανίζουν, αλλά μου λένε έχουμε τόσο πολλούς ελέγχους, δεν, έχουμε καν, δεν θέλουμε καν να κάνουμε αίτηση γιατί όλο ελεγκτές έρχονται και τα λοιπά. Γι' αυτό ακριβώς προσπαθούμε να έχουμε μια αξιοπιστία στον ε, έλεγχο, να σεβαστούμε και την αρχή της επικουρικότητας και να ρυθμιστεί αυτό στο πρώτο επίπεδο γιατί κάπου πρέπει να αντιληφθούμε πως ε, πρέπει να υπάρχει μία κάποια ισορροπία. Και αν υπάρχει μια αξιοπιστία, όπου υπάρχει μια αξιοπιστία του ελέγχου, τον εμπιστευόμαστε. Τώρα για τις αιτήσεις δραστηριότητες, όπου έχουμε μια ένδειξη πως δεν λειτουργούν τα προγράμματα, αμέσως προχωράμε σε διακοπή. Εισηγητής θα ήθελε να κάνει κάποια καταληκτικά σχόλια. Η κυρία Γιάλα Σέντερ. Α, σας ξέχασα, δεν θα γίνεται αριστερά. Συγγνώμη, πρόεδρε. Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Χάν. Γίνονται διορθώσεις, έγιναν διορθώσεις μάλλον στην περίοδο 2000-2006. Ξέρω ότι έκανα πολλές ερωτήσεις, δεν απαντήσατε όμως σε αυτή την ερώτηση. Ε, ο κύριος Πίπερ νομίζω φτάνει σε λανθασμένα συμπεράσματα. Ε, το 2000-2006 για την Ισπανία έγιναν διορθώσεις. 1.800 ε, δις. Αυτό το ποσό έχει ήδη διορθωθεί πριν το 2010. Τώρα άλλαξαν οι λογιστικοί κανόνες και το ξαναυπολογίζεται και ξαναυπολογίζεται όλη αυτή τη διόρθωση. Δηλαδή το 2012 έγινε διπλή διόρθωση. Είχε γίνει ούτως ή άλλω η αλλω η μία φορά πριν το 2010 και ξανά έγινε μετά. Εγώ δεν το λέω. Δεν το λέω εγώ αυτό. Είναι γραμμένο αυτό που σας λέω. Δεν το επινόησα. Αρκεί να διαβάσετε τις υποσημειώσεις που μιλάμε για τη συνολική διόρθωση για την Ισπανία, την καθαρή διόρθωση, είναι 1,8 δις. Και οφείλεται στο γεγονός ότι γίνεται ως υπολογισμός της διόρθωσης. Μία φορά έγινε το 2006 ας πούμε και τώρα ακόμα μία φορά γιατί κλείνει αυτή η περίοδος. Κλείνουν τα βιβλία για αυτή την περίοδο. <clears throat> Δεν θέλω να βάζετε μόνιμα στην Ισπανία στους ε, κακούς μαθητές, ε, κύριε Πίπερ, έτσι. Σύντομα. Ε, μιλήσαμε για την περίοδο 2000 με 2006, έτσι, και το θέμα είναι πως το 2012 μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις για τις δημοσιονομικές διορθώσεις σε μεμονωμένα έργα της περίοδου 2000-2006. Και στην περίοδο 2000-2006 έπρεπε κάθε έργο να ε, υπολογιστεί. Όχι πρόγραμμα, αναέργο, έτσι, να γίνει απολογισμός. Και είχαμε συζητήσεις με τις διάφορες ισπανικές κυβερνήσεις για τις δημοσιονομικές αυτές διορθώσεις και η προηγούμενες ισπανικές κυβερνήσεις ήθελαν να συζητηθεί κάθε έργο μέχρι το τέλος. Εννοούσαν δηλαδή μέχρι και το ΔΕΚ. Έτσι. Και καταλήξαμε σε μία συμφωνία με την ε, κυβέρνηση, την ε, τωρινή, για τις δημοσιονομικές διορθώσεις, για όλα τα έργα, εφαρμόστηκε σε όλα τα έργα, κατά το οποίο οδήγησε στο ότι το 2012 έκλεισε αυτό το ζήτημα και ε, πρόκειται ακριβώς για πολύ υψηλές δημοσιονομικές διορθώσεις άπαξ οι οποίες καλύπτουν την περίοδο 2000-2006 και έκλεισαν σε ένα χρόνο. Κάτι το οποίο βεβαίως είχε ως αποτέλεσμα το 2012 όσον αφορά τον ε, ισπανικό προϋπολογισμό ε, είχαμε ε, κάποια μείωση του ισπανικού προϋπολογισμού αλλά είχαμε νομίζω ούτως ή άλλως γύρω στο 1 δισεκατομμύριο χρηματοδότηση. Οπότε έτσι έχουν τα πράγματα, ούτως ή άλλως δεν προκαλεί και καλή εντύπωση το να μην μπορούμε να κλείσουμε τα βιβλία του 2000-2006. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Πίπερ θα ήθελε να ολοκληρώσει. Ναι. Ε, μετά από αυτό το διάλογο νομίζω πως χρειαζόμαστε οπωσδήποτε έκθεση για την Ισπανία τουλάχιστον, έτσι. Και θα πάρουμε μόνο μία Ισπανική περιφέρεια και τη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία, έτσι και στις δύο περιπτώσεις περιφέρειες και στις δύο περιπτώσεις ε, ομοσπονδιακή δομή και ελπίζουμε πράγματι ε, να σκεφτείτε αυτό το οποίο είπαμε. Είναι κάποια, αυτά είναι κάποια από αυτά τα οποία είπατε ενθαρρυντικά. Αυτό για το οποίο ακούστηκε πως δεν μπορεί ε, να τα κάνει αυτά κάθε χρόνο το ελεγκτικό συνέδριο δεν το ζητάμε. Δύο-τρεις χώρες κάθε χρόνο, ένα λάξ. Έτσι νομίζω αυτό είναι εντό των δυνατοτήτων του. Έμαθα πολλά πράγματα σήμερα και οφείλω να πω πως ε, γενικά η εντύπωση είναι θετική. Τώρα πολλά θα εξαρτηθούν από τις επόμενες εβδομάδες. Αυτό το οποίο... Α, δεν ε, βλέπω εγώ και δεν μπορώ να παρακολουθήσω είναι το πώς θα μπείτε στην διαδικασία αυτή, το πώς ξεκινάει αυτή η διαδικασία ελέγχου. Δηλαδή ότι όταν ξεπεράσουν το 2% τα κράτη-μέλη παρεμβαίνει η Κομισιόν. Δεν μου φτάνει. Εγώ θα ήθελα κάποια κριτήρια τα οποία θα είναι, ξέρω εγώ, αυτό ανέλησε στο παρελθόν το ελεγκτικό συνέδριο. Είχαμε και ένα δειγματοληπτικό έβριμα της ε, Κομισιόν, συν ε, υπέρβαση του 2%, δηλαδή κάποια κριτήρια σωρευτικά με τα οποία λέμε από εκεί και πέρα παρεμβαίνουμε. Τέλος, κύριε Επίτροπε, 700 υπάλληλοι από τους οποίους 83 ε, στον έλεγχο. Δεν είναι πολύ. Είναι τρομακτικό δηλαδή το πόσοι λίγοι ασχολούνται πανευρωπαϊκά με τον έλεγχο. Ναι, στη Γενική Διεύθυνση, ναι. 83 για τόσα πολλά προγράμματα και έργα δεν είναι πολύ. Αν δούμε το τι έχουν άλλες γενικές διευθύνσεις ε, και το τι παράγουν έτσι ως ευρωπαϊκή Προστασία δεν θέλω τώρα να κατονομάσω, αλλά θα μπορούσε να υπάρξει μια αύξηση νομίζω του προσωπικού. Αναμένω λοιπόν το τι θα ακολουθήσει επόμενες εβδομάδες και τη συνεργασία μας. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι τελείωσε αυτό το σημείο της μέσης διάταξης. Μάλλον κάνατε μεγάλη εντύπωση με την ομιλία σας. Θα θέλαμε να, την, να, μας τη στείλετε. Θα μας τη στείλετε φαντάζομαι στα γερμανικά. Σας ευχαριστούμε Επίτροπε. Ευχαριστούμε τον κύριο Γκρέτεν. Και τώρα περνάμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης. Sorry? Voting list? I have the voting list here. We can just start. Yeah.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 Okay, okay. Okay. Nou ja, okay. Okay, niks eraan te doen. Hartstikke Dank. Είστε έτοιμοι για να αρχίσουμε την ψηφοφορία. Okay. No problem. I suggest we... Προτείνω λοιπόν να ξεκινήσουμε. Έχουν όλοι την κάρτα τους για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Then I open the vote. Εάν ναι, μπορούμε να ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία επί του σχεδίου γνωματότησης για το διαδικασία διορισμού των μελών του ηλεκτρικού συνεδρίου και την διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξεκινούμε με το 13, τροπολογία 13, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 14, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 15, υπέρ. 15, 15. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος καλύτερα. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Πρέπει να πατήσετε το κουμπί, λέει ο Πρόεδρος. Ωραία, πέρας ψηφοφορίας. Ε, ε, Δέκα υπέρ, οκτώ κατά. Σύνολο 18 ψήφι. Καμία αποχή. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17 αποκαταπίπτει, το ίδιο και η 16. Παρακαλώ. Για την ακρίβεια το αποτέλεσμα είναι σωστό, αλλά νομίζω πως ε, οι Ίνες ε, ήταν κατά έτσι και είναι ναι. Ναι, αλλά πάλι εγκρίνεται. Amendment 17 false. Amendment 16. Καταπίπτουν οι τροπολογίες 16 και 17 και τώρα ψηφίζουμε για την 18. Υπέρ 18. Κατά. καλύτερα να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο έναρξης ψηφοφορίας. Πέρας. 12 υπέρ, 7 κατά, εγκρίνεται. Προπολογή 19, υπέρ. Κατά. κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο γιατί δεν σηκώνετε αρκετά ψηλά το χέρι σα. Ε, Έναρξη ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Και έχουμε ισοψηφία. Και απορρίπτεται. 9 υπέρ, 9 κατά, απορρίπτεται. Ε, τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ε, ρωτά πρόεδρο, υπάρχουν αποχέ, όχι εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ. Θέτω στη ψηφορία την 21 γιατί η 19 δεν εγκρίθηκε. 21 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 22. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Το ε, συγγνώμη δεν υπήρχαν αποχές. Ωραία εγκρίνεται. λέγει 23. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. λέγει 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1, η οποία αντικαθιστά τις 26 έως 28. Ποιος είναι υπέρ συμβαστικής 1, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τρόπο 25, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Καταπέπτουν 26, 7 και 8. Τροπολογία 29. Υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορριφθήκε, αλλά στο ελέγξουμε. Έναρξη ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρα. 9 υπέρ, 10 κατά, απορρίπτωται. Τροπολογία 30 υπέρ. Αποχές. Εγκρίνεται. 31 καταπίπτει. Τροπολογία 32. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος, ηλεκτρονική ψηφορία, παρακαλώ ψηφίστε. Πέρασε. Εγκρίνεται με 10 ψήφους υπέρ 9 κατά. Καταπίπτει 33, σωστά. Το ίδιο και η τροπολογία 34 και, και αυτή καταπίπτει. Και πηγαίνουμε στην συμβιβαστική νούμερο 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. που σημαίνει ότι καταπίπτουν οι 35, 36 και 37. Τροπολογία 38 υπέρ. Κατά. Ας κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Έναρξη ψηφορίας. Πέρας. Ισοψηφία 10 υπέρ 10 κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 39 υπέρ. Κατά. Νομίζω πως συγκρίνεται. Τροπολογία 40 υπέρ. Κατά. Ας το ελέγξουμε. Έναρξη ψηφορίας. Πέρας mm. Και πράγματι απορρίπτεται. Τροπολογία 41 υπέρ. Κατά. Ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 42. Υπέρ. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά αμέσως αμέσως έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Άρα καταπίπτουν οι 43, 44 και 45. Τροπολογία 46. Ποιος είναι ε, υπέρ. Και η τροπολογία 47 είναι η ίδια. 46 ή 47 υπέρ. Κατά. Νομίζω πως εγκρίνεται. Τροπολογία 48 καταπίπτει, το ίδιο και η 49 και πηγαίνουμε στην τροπολογία 50. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία νούμερο 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. που σημαίνει ότι καταπίπτουν οι 53, 54 και 55. Και 52. Και προχωρούμε στην τροπολογία 56. 56 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 57 και 58 καταπίπτων. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Έναρξη. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 59 καταπίπτει το ίδιο και η 60, το ίδιο και η 61. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 62, 62 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 63 υπέρ. Δεν μπορώ να το ξεχωρίσω για να χειρός. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία, 13 υπέρ, 7 κατά. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 64 έχει αποσυρθεί, 65 κατά πίπτη. Τροπολογία 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 67. υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορίας για τη συμβιβαστική 5. Ψηφίστε. Πέρας ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. Που σημαίνει ότι θα χρειαστεί να ψηφίσουμε ξεχωριστά ε, πρώτα απ' όλα την 68. Σωστά. Ναι. Τροπολογία 68 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 69. Υπέρ. Αφού η συμβιβαστική 5 δεν εγκρίθηκε, πρέπει να ψηφίσουμε ξεχωριστά τις υπόλοιπες τροπολογίες, λέει ο πρόεδρος. Α, λάθος. Συγγνώμη, διορθώνει ο πρόεδρος. Στην 73 έπρεπε να πάμε. Τροπολογία 73. Εδώ υπάρχει προφορική τροπολογία που μπορείτε να αναγνώσετε στον κατάλληλο ψηφοφορίας. 73 υπέρ. Καλύτερα να το θέσω κατευθείαν σε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Παρακαλώ ψηφίστε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 74. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 74 εγκρίθηκε, πράγμα που σημαίνει ότι καταπίπτει η 75. Και η 76. Αλλά όχι, για την 76 πρέπει να ψηφίσουμε. 76 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία τα ε, και 78 και 79 καταπίπτουν. Τροπολογία 80 υπέρ. Κατευθείαν ηλεκτρονικό έλεγχο προτείνω. Έναρξη της για την 80. περε ψηφοφορια ψηφοφορίας. 10-11. Ε, απορρίψετε. Τροπολογία 81. 81 υπέρ. ηλεκτρονικά κατευθείαν. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. Για δες, εγκρίνεται. Έχει αποσυρθεί 82, η 83 καταπίπτει, το ίδιο και η 84 και προχωρούμε με τη συμβιβαστική τροπολογία 6. Συμβιβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Που σημαίνει Το πρώτο μέρος της 85 καταπίπτει, αλλά θα πρέπει να ψηφίσουμε για το δεύτερο μέρος. Δηλαδή τη διαγραφή από το emphasizes μέχρι το τέλος. πρέπει να ψηφίσουμε για το δεύτερο μέρος της 85 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 86-87 καταπίπτουν. Τροπολογία 88 υπέρ. Αποχές, ε, συγγνώμη, ε, κατά πρώτα απ' όλα. Ποιος είναι κατά στην 88. Αποχέ. τώρα. Απορρίπτεται. Η 89... Ε, όχι, με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρο την 89 πρέπει να την ψηφίσουμε, γιατί 88 δεν εγκρίθηκε. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 90 έχει αποσυρθεί. Τροπολογία 91 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 93 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 95. 95 υπέρ. 95. Θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζετε τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 96 Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 97. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 98. Υπέρ. Θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 99. Πρέπει να ψηφίσουμε σε δύο τμήματα. Αυτή είναι η τροπολογία υπέρ του πρώτου τμήματος, κατά, αποχές, εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά. Νομίζω ότι περισσότερο είναι υπέρ, αλλά στο τσεκάρουμε. Ψηφίστε ηλεκτρονικά. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 99. Πέρας φοφορίας. Απορρίπτεται. 100. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 101 υπέρ κατά δεν είναι σαφές ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τώρα την 101 πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται θα ελέγξουμε την 103 ηλεκτρονικά The vote is closed. Πέρας προφορίας 15 υπέρ 6 εποχές. 104 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ. Κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται. 106 Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 107. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 108. Υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας προφορίας. Εγκρίνεται. 109 με προφορική τροπολογία που αλλάζει μια λέξη. Το explores το κάνει deplores. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. στα ισπανικά το κείμενο για αυτή την τροπολογία έχει πρόβλημα. Πέρα από το explores, deplores, το βασικό είναι να ονομάζουμε σωστά και τις, τα γραφεία των επιτρόπων. Να μην λέμε το καμπινέ των επιτρόπων, να λέμε το γραφείο των επιτρόπων, έτσι, στα ισπανικά, έλεος. Ναι, ναι, θα ζητήσω από τι αρμόδιε υπηρεσίε να το διορθώσουν. Εγώ δεν μπορώ να σα βοηθήσω με την ισπανική μετάφραση, αλλά το καταγράψαμε. 110. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 111. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η μία ομάδα της αίθουσας αδιαφορεί πλήρως για αυτό το σημείο. Για να το ψηφίσουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Α, εγώ το, το υποπτευόμουν, αλλά οι υπόλοιποι δεν ήταν σίγουροι. Αυτό σημαίνει ότι 113, 114, 115 καταπίπτουν και πάμε στην 116. Υπέρ της 116 με την προφορική τροπολογία όπως βλέπετε στο κείμενό σας. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 117. Υπέρ, κατά. Δύσκολο να το καταλάβω. Για να το δούμε ηλεκτρονικά παρακαλώ ψηφίζετε τώρα. Πέρας φοφορίας. Απορρίπτεται. 118 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 119 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά στο τσεκάρουμε ηλεκτρονικά. Το 119. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 120 καταπίπτει. Συμβαστική τροπολογία 8. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 122, 121 και 123 ψηφίστε τώρα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 124 μέχρι υπέρ. Ψηφίζουμε την 124 και 125 που είναι οι ίδιες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 126 υπέρ. Ψηφίζουμε την 126, δεν καταπίπτει. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά στο επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε τώρα. τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 128. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 129. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 130. Υπέρ. Κατά. Δεν ξέρω. Επαληθεύουμε τώρα το σημείο αυτό ηλεκτρονικά. Ψηφίζεται. Πέρας φοφορίας. Εγκρίνεται. 131 falls. 131 καταπίπτει. 132. Ψηφίσουμε τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 132. Λέει ο Πρόεδρος. Διορθώνει όχι, δεν ήταν σωστό. Την 133 εννοεί. Την 132 την ψηφίσαμε. Πάμε στην 133 λοιπόν και 134 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για αυτές τις δύο. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 135 κατά πίπτη. 136 και 137. Υπέρ παρακαλώ. Για θέσεις 2. Κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε τώρα. Πέρα σχοφορίας. Εγκρίθηκε. 138 λοιπόν καταπίπτει. Ψηφίσουμε την 139 και 140 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται νομίζω. Η 141 λοιπόν καταπίπτει και η 142. Ψηφίσουμε τα 143 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι περισσότερο είναι υπέρ, αλλά ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρα φοφορίας. Απορρίπτεται. 144 υπέρ. Κατά. Yes. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 145 και 146 λοιπόν. Υπέρ των δύο αυτών τροπολογιών. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 147. Καταπίπτει. 148 καταπίπτει. Και πάμε στην 149. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 150. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 151. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 152. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 153. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίθηκε. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 155 κατά αποχές απορρίπτεται 156 υπέρ κατά εγκρίνεται η 157 καταπίπτει 158 ψηφίζουμε υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται το 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 162 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 163 υπέρ δεν καταπείτε. την ψηφίζουμε υπέρ της 163 κατά αποχές εγκρίνεται 164 υπέρ κατά δύσκολο να καταλάβω ηλεκτρονική επαλήθευση ψηφίστε τώρα πέρα ψηφοφορίας εγκρίθηκε 165 υπέρ κατά η ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζεται τώρα. Πέρας. Απορρίπτεται. 166 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται. 167 κατά πίπτη. 168 υπέρ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 169 κατά πίπτη. Υπέρ της 170. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 171 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 172 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 173. Κατά εποχές απορρίπτεται. 174 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 175 υπέρ ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίστε τώρα. Πέρας φοφορίας. Απορρίφθηκε. Πρώτη τροπολογία. Και δεύτερη. Ένα και δύο. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνονται. Τρία. Προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Άποχες. εγκρίνονται Τέσσερα. Υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 σε δύο τμήματα ε, πρώτο τμήμα υπέρ του πρώτου τμήματος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά δεν σαφές ηλεκτρονική επαλήθευση ψηφίστε τώρα πέρα φοφορίας Εγκρίνεται. 11. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε στο ψήφισμα συνολικά όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε τώρα. Πέρας ψηφοφορία. Απίστευτο αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. I hope she is as happy as we are. Ελπίζω να είναι και εκείνη τόσο ευτυχής όσο και εμείς. Πάμε στην επόμενη ψηφοφορία. Εκτός μικροφώνου. Κανείς θα παραπονεθεί για το θέμα της δομής του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου. Πήραν αυτό που ήθελαν και ελπίζω τουλάχιστον εκείνοι να μην παραπονεθούν. Δεν μπορώ να ακούω άλλα παράπονα. Βαρέθηκα τα παράπονα. Πάμε στην δεύτερη έκθεση, σχέδιο γνωμοδότησης για ένα κανονισμό του Συμβουλίου για το ECSEL, την κοινή επιχείρηση αυτή. Ψηφίζουμε κατευθείαν. Ο εισηγητής να πει δυο λόγια. Νομίζω μπορούμε να ψηφίσουμε το 1 ως 17 μπλοκ. Συμφωνούν όλοι. Ωραία. Τίθεται σε ψηφοφορία. Από το 12 μέχρι το 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Γιατί εγκρίνονται. 18. Υπέρ. Κατά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τώρα. The vote is closed. Πέρας Απορρίφθηκε. 19. για 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Νομίζω δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε την 20, ρωτά ο πρόεδρος. Όχι, όχι, λάθος. Πρέπει να ψηφίσουμε την 20. 20 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασε. Εκρίνεται, που σημαίνει ότι καταπλήττει η τροπολογία 1. Και τώρα ψηφίζουμε για την 21. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 22. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 23. Υπέρ. Ας ελέγξουμε κατευθείαν ηλεκτρονικά έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Που σημαίνει ότι καταπίπτει 2 και μπορούμε να ψηφίσουμε την 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 25 υπέρ. Εντελώ ασαφές ηλεκτρονικός έλεγχος λοιπόν, ε, έναρξη ψηφοφορίας, πέρασε. Εγκρίνεται που σημαίνει ότι καταπίπτει η 3 και μπορούμε να ψηφίσουμε την 26. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ. Κατά Εγκρίνεται. Όχι, όχι, ας ελέγξουμε καλύτερα. Έναρξη ψηφοφορία για την τροπολογία 27. Πέρας ψηφοφορίας. Ευτυχώς που ελέγξαμε. Ε, η ισοψηφία 9-9 ναι, που σημαίνει ότι απορρίπτεται. 28. Υπέρ. Ας, ας περάσουμε κατευθείαν σε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. 17. Εγκρίνεται. Τροπολογία 29. Υπέρ. Ηλεκτρονικά κατευθείαν. Παρακαλώ ψηφίστε. Πέρας ψηφοφορία. 8 υπέρ, 9 κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Λάθος. Ε, συμβιβαστική τροπολογία μάλλον. Συμβιβαστική. Υπέρ. Κατά. Αποχές, καμία, επομένως εγκρίνεται. Εγκρίνεται η συμβαστική τροπολογία 1. Αυτό δεν έχει καμία επίπτωση όμως στις υπόλοιπες. Πρέπει να συνεννοηθούν εδώ πέρα νομίζω οι συνάδελφοι, οι δύο συνάδελφοι του ΕΛΚ έτσι έρχονται. Όχι, όχι. Εντάξει, Ρούμπιχ και Ουντί πρέπει να, να συνεννοηθούν. Ε, ναι. Πλησιάζουν και τα Χριστούγεννα και θα συνεχίσουμε σε αυτό το κλίμα να ψηφίσουμε. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ. 7 Αποχές. Εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8 αποσύρεται. Αν έχω καταλάβει καλά. 9 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 35 σε δύο μέρη μέρος πρώτο υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται μέρος δεύτερο υπέρ κατά Α, εγκρίνεται τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές αντεκτή 36 υπέρ κατά ε, δεν είναι σαφές ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται πέρας δεκτή 37 υπέρ 37 και 38 μαζί υπάρχει αντίρρηση όχι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 39 υπέρ αντιρρήσει για να ψηφίσουμε 39 40 μαζί, όχι. 39-40 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται και οι δύο. 41 υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές. Θα ψηφίσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 43 με 48 αμπλοκ αντιρρήσεις. Ορίστε. 43 και 44. Υπέρ. Κατά. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 45. Υπέρ. Κατά. Νομίζω πως η φιλοψηφία είναι υπέρ. 48 ποιος είναι υπέρ 47-46 πίπεν κατά δεν είναι σαφές ηλεκτρονική ψηφοφορία αρχιετή ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές δεκτή 50 υπέρ κατά δεν είναι σαφές. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρασε. Δεκτή. Τροπολογία 51 υπέρ. Ναι, όλα μαζί. 51 έως 56. Υπάρχει αντίρρηση, όχι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται όλες περνάμε στην τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία πέρας συγχαρητήρια στον εισηγητή με συντριπτική πλειοψηφία διακόπτουμε για δύο λεπτάκια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

με την άδειά σας. Να συνεχίσουμε την ημερήσια διάταξη. Και περνάμε στο σημείο 7, την ειδική έκθεση, νούμερο 5 του 2013, για την πολιτική συνοχής. Χρησιμοποιούνται σωστά οι πόροι για τους οδικούς άξονες. Ο κύριος Βέγκερ Πάουερ πρώτα απ' όλα. Έχετε το λόγο. Και σας ζητώ να μην μακρηγορήσετε. γιατί ήταν κάπως φορτωμένη η ημερησία μας διάταξη απόψε. Είμαι σύντομος. Χαίρομαι για το ότι υπάρχει τόσο πολύ ενδιαφέρον για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Τώρα περνάμε στα συγκεκριμένα από την δήλωση αξιοπιστίας. Θα προσπαθήσω λοιπόν να είμαι σύντομος. Το ερώτημα είναι εάν τα κονδύλια ε, που διατίθενται για τα οδικά δίκτυα αξιοποιούνται ορθά. Διαπιστώσαμε δύο πράγματα. Μεγάλες διαφορές κόστους στους δρόμους που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συχνά έχουμε ακριβούς δρόμους και όχι αποτελεσματικούς ως προς το κόστος. Γιατί και πώς είναι το αντικείμενο της έρευνάς μας. Οι επενδύσεις στα οδικά έργα κάθε χρόνο είναι γύρω στα 5 δισεκατομμύρια το έτος. Εξετάσαμε 24 ε, έργα σε Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία και Πολωνία. Για αυτά τα έργα έδωσε γύρω στο 1,4 δισεκατομμύριο ε, αναέργο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γύρω στο 62% δηλαδή ήταν η συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 62% ε, της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τις χώρες αυτές 2000 ε, με 2013. Πρώτη βασική διαπίστωση, μεγάλες διαφορές κόστους. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αξιολόγησε με τρεις τρόπους υπολογισμού το κόστος για να μην μπορεί κανείς να πει πως πήραμε κάποια στοιχεία αποσπασματικά για ένα έργο ή ένα κράτος. Και με τους τρεις τρόπους υπολογισμού ήταν πιο φτηνή η γερμανική δρόμη και μετά κατά σειρά Ελλάδα, Πολωνία και Ισπανία. Η Ισπανία και με τους τρεις τρόπους υπολογισμού ήταν δύο φορές πιο ακριβή από τη Γερμανία. Εάν το δούμε με την ένταση χρήσης, η ε, ισπανική δρόμη είναι τέσσερις φορές πιο ακριβή από τους γερμανικούς και βέβαια το ερώτημα είναι πώς γίνεται. Εργασιακό κόστος ε, δεν μπορεί να είναι η διαφορά γιατί δεν είναι και τόσο φτηνά τα εργατικά στη Γερμανία. Οπότε ποιες είναι οι πιθανές εξηγήσει. Πρόκειται για ε, θέμα ανταγωνισμού. Ε, στην ε, Γερμανία είχαμε μικρούς διαγωνισμούς λίγων χιλιόμετρων, ένα-ενάμιση, ενώ στις υπόλοιπες χώρες είχαμε δημοπράτηση μεγάλων έργων στη Γερμανία και στην Πολωνία μπορούσαν να συμμετέχουν όλες οι εταιρείες. Σε Ελλάδα και Ισπανία όχι. Εδώ πέρα έπρεπε να υπάρχει μια πιστοποίηση πρώτα από τις ε, δημόσιες αρχές, κάτι το οποίο βέβαιως επηρέασε τον ανταγωνισμό και σημαίνει μεγάλο διοικητικό άχθος το οποίο οδηγεί και σε καθυστέρηση της πιστοποίησης αυτής. Στην Ισπανία και στην Ελλάδα έγιναν προσφορές κατά 10% μικρότερες από το μέσο... Ε, αυτές οι οποίες ήταν κατά 10% μικρότερες από το μέσο κόστος αποκλείστηκαν. Οι Κομισιόν βεβαίως αντέδρασε με ένα πρόστιμο 10% το οποίο βεβαίως οδήγησε στο ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες αποκλείστηκαν με αυτό τον τρόπο αργότερα έκαναν κοινοπραξίες με αυτούς οι οποίοι κέρδισαν τον ε, διαγωνισμό. Τέταρτον, για, το για τη διαφορά του κόστους, το τείχος προστασίας ε, του θορύβου έπρεπε ε, να είναι υπερβολικών διαστάσεων ε, στην Πολωνία λόγω εθνικών διατάξεων. Εάν πάει κανείς σε αυτοκινητόδρομο στην ε, Πολωνία δεν βλέπει καθόλου τοπίο, μόνο το τείχος αυτό προστασίας του από τον θόρυβο. Επίσης, πέμπτο, υπήρχε μεγάλη διαφορά κόστους και σε άλλα κριτήρια εξοπλισμού όπως πινακίδες κτλ. Και εκεί πέρα είχαμε κάποιες διατάξεις ε, οι οποίες στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, οι οποίες πρέπει να παραμεριστούν, γιατί σημαντικότερος, ε, σημαντικός ε, στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης βεβαίω είναι η ενίσχυση του ανταγωνισμού. Οπότε, πρώτο, απέτηση από τον Επίτροπο Ανταγωνισμού να υπάρχει συνολικός ανταγωνισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να υπάρχουν οι δυνατότητες να αρθούν όλα τα εμπόδια στον ανταγωνισμό. Επίσης, κάτι άλλο. Σε όλα τα έργα τα οποία εξετάσαμε, βρήκαμε μόνο ένα έργο το οποίο ε, ανέλαβε ξένη εταιρεία. Αυτό δείχνει πως πρέπει να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα, η η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Αυτή είναι η βασική μας απέτηση από τον Επίτροπο Ανταγωνισμού. Αυτό σημαίνει έρευνα των ενιών, των ε, αιτιών με συγχωρείτε, για τις μεγάλες αυτές διαφορές του κόστους ε, στην καταστροφή, στην κατασκευή δρόμων και βεβαίως ε, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτών. Δεύτερον, όπως είπα, να παραμεριστούν τα εμπόδια στον εσωτερικό ανταγωνισμό. Τα ανέφερα ήδη το ποιοι ήταν οι ανάδοχοι των έργων και πάρα πολλά έργα μπορούσαν να τα αναλάβουν μόνο μεγάλες επιχειρήσεις ε, λόγω των ε, όρων του διαγωνισμού γιατί όπως είπα προκυρήσονταν ε, 250-500 χιλιόμετρα τη φορά και τίθεται και το ζήτημα της ε, πιστοποίησης των εταιριών. Δεύτερο, που θέλουμε να αναφέρουμε, έχουμε ακριβούς ε, δρόμους αντί για έργα τα οποία θα ήταν πιο αποτελεσματικά ως προς το κόστος και τις ανάγκες. Μετά είδαμε πως το μέσο κόστος για δρόμους ε, ταχείας κυκλοφορίας είναι κατά 53% πιο φθηνή από τους αυτοκινητόδρομους. Τώρα, τους χρειαζόμαστε τους αυτοκινητόδρομους ή όχι. Κοιτάξτε, βλέπουμε μια χρήση η οποία κυμαίνεται στους μεν δρόμου από 16.900 ημερησίω ενώ στην άλλη περίπτωση 13.390. Οπότε το ακριβότερο δεν σημαίνει οπωσδήποτε καλύτερο. Σε πάρα πολλές ε, περιπτώσεις ε, νομίζω πως ε, η απλή δρόμη ταχεία κυκλοφορία είναι η καλύτερη και οικονομικότερη λύση. Γιατί λοιπόν έργα τόσο μεγάλων διαστάσεων. Οι αιτίες είναι οι πάρα πολύ αισιόδοξε εκτιμήσεις για την ε, κίνηση, για την κυκλοφορία. Αυτό οδήγησε στο ότι το μέσο κόστος ε, ενός χιλιόμετρου δρόμου σε σύγκριση με την ε, κυκλοφορία που περνάει από εκεί σε ένα έτος στην ε, Ισπανία ήταν ε, τέσσερι φορές μεγαλύτερο από ό,τι στη Γερμανία. Πολωνία και Ελλάδα ήταν στη μέση μεταξύ των δύο άκρων. Οπότε τίθεται το ζήτημα πώ οδηγούμαστε σε τόσο υπεραισιόδοξε προβλέψει, Είναι και πολιτικό βεβαίω το ζήτημα το οποίο δεν θα κρίνουμε εμεί, αλλά είναι σαφές ε, πως αυτό πρέπει να το κάνουν τα κράτη-μέλη σε συνεργασία με την Κομισιόν. Ε, το κόστος ε, αναχρήστη ε, παρουσιάζει μια ψαλίδα που είναι και 28 φορές μεγαλύτερη. Το υψηλότερο με το χαμηλότερο. Και βεβαίως, όπως είπαμε, είχαμε καθυστερήσεις μέχρι και ε, νέα μήνες οι οποίες οδηγούν σε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση του κόστους. Και βεβαίως ε, τίθετο το ζήτημα όπως είπα των αξιόπιστων προβλέψεων της ε, κίνησης. Εδώ πέρα διαπιστώσαμε με ευχαρίστηση πως η Κομισιόν κάτι ήδη έχει κάνει και όσον αφορά βεβαίως και τις υπερβολικές απαιτήσει όσον αφορά τα έργα διαφορών κρατών μελών τα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες, στις πραγματικές. Θα ήθελα μετά από αυτά τα οποία είπα να κλείσω με κάτι το θετικό αφού ανέφερα τα βασικά σημεία κριτικής. Διαπιστώνουμε πως η βασική στόχη, δηλαδή καλύτερη διασύνδεση των περιφερειών, καλύτερη οδική ασφάλεια, καλύτερη άνεση κτλ, ενίσχυση των υποδομών, επιδέχθηκαν. Το πρόβλημα το οποίο έχουμε εδώ πέρα είναι βεβαίως η ενίσχυση των υποδομών η οποία πρέπει να μετρηθεί. Γι' αυτό πρέπει εδώ πέρα η Κομισιόν να ε, δώσει μια συνέχεια, δηλαδή να δει εάν τα μέτρα αυτά υποδομών είναι θετικά μεσομακροπρόθεσμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο εισηγητής, θα ήθελα να αντιδράσει σε αυτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο και το μέλος υπεύθυνο για την εκπόνηση της έκθεσης, τον κύριο Χάραλαντ Μπάουερ για την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση που μας παρουσίασε και την εξωτερική συνεργασία που είχαμε. Καταρχήν θα ήθελα να καλωσορίσω τα ευρήματα του Ελεκτικού Συνεδρίου που επιβεβαιώνουν ότι έχει υπάρξει μια αξιοσημείωτη βελτίωση στην οδική ασφάλεια και μια σημαντική μείωση των θανάτων στην άσφαλτο. Μάλιστα, σε μερικέ περιπτώσει έχουμε μηδενικό αριθμό θανάτων που βελτιώνουν την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στα μεγάλα έργα υποδομή και έχουν θετικό αντίκτυπο στα δημόσια οικονομικά του, στου τομεί τη δημόσια ασφάλεια και τη δημόσια υγεία. Θα ήθελα επίση να καλωσορίσω το γεγονό ότι το συνέδριο συμπέρανε ότι υπήρξε μείωση στον χρόνο ταξιδίων και σε σύγκριση με εναλλακτικέ συγκοινωνιακέ συνδέσει υπήρξε εξοικονόμηση χρόνου έως και 60%. Είμαι πεπισμένο ότι οι παραπάνω βελτιώσει θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία και μπορούν να δημιουργήσουν νέε θέσει απασχόλησης. Είναι σημαντικό το ότι για αυτά τα οδικά έργα είχαν τεθεί στόχοι όσον αφορά τα αναμενόμενα αποτελέσματα Ωστόσο, ο αντίκτυπος που είχαν τα έργα αυτά στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας ή η πραγματική ωφέλεια για τους χρήστες του οδικού δικτύου δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθεί εξαιτία της έλλειψης κατάλληλων δικτών. Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περίοδου θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν ένα αξιόπιστο και μετρήσιμο αριθμό δικτών προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό. Επιπλέον, θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο η Επιτροπή να συνεχίσει να ανανεώνει και να προσαρμόζει τον οδηγό που έχει εκδώσει σχετικά με την ανάλυση κόστος-οφέλους των επενδυτικών έργων και να παρέχει καθοδήγηση για τι προβλέψει όσον αφορά την κυκλοφορία στα δικά έργα. Επίση, κάνω έπειση στην Επιτροπή να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών με σκοπό από τη μία μεριά να υπάρξουν αξιόπιστε κυκλοφοριακέ προβλέψει και από την άλλη να υπολογιστεί ο πιθανό οικονομικό αντίκτυπο των οδικών κατασκευών. Όσον αφορά το κόστο τη κατασκευή δρόμων, είμαι τη άποψη ότι εξαρτάται από πολλού παράγοντε όπω η μορφολογία του εδάφου, η τοπογραφία, η σεισμική επικινδυνότητα, η περιβαλλοντική, η αρχαιολογική και πολιτιστική περιορισμοί που υφίστανται, καθώ και από τα συμπληρωματικά τεχνικά έργα που απαιτούνται για την κατασκευή των δρόμων, όπω για παράδειγμα γέφυρε και σύραγγες. Πρόκειται να σα δώσω ένα παράδειγμα για το τι συμβαίνει στη χώρα μου, λαμβάνοντα υπόψη για την επιστημονική μου εμπειρία. Η Ελλάδα είναι η πλέον σεισμογενή χώρα τη Ευρώπη και η πέμπτη στον κόσμο. Το 90% τη σεισμική ενέργεια απελευθερώνεται στην Ελλάδα σε σύνολο τη Ευρώπη. Ισχυροί σεισμοί με μέγεθο μεγαλύτερο του 5,5 βαθμών τη κλίμακα Ρίχτερ συμβαίνουν συχνά με μέση περίοδο επανάληψη περίπου 6 μηνών. Όλε οι κατασκευέ σχεδιάζονται σύμφωνα με τον αυστηρό εθνικό αντισυσμικό κανονισμό και τον Ευρωκώδικα νούμερο 8. Κρίσιμε κατασκευέ όπω αγωγή φυσικού αερίου, γέφυρε, φράγματα, σύραγγε, οδικοί άξονες κλπ. Σχεδιάζονται με αυστηρά κριτήρια λαμβάνοντα υπόψη τι τοπικέ εδαφικέ συνθήκε, την πιθανότητα κατολιστήσεων, καταπτώσεων βράχων, ρευστοποίηση του εδάφου κλπ. Ειδικότερα γραμμικά έργα όπω παραδείγματο χάρη αγωγή φυσικού αερίου, αυτοκινητόδρομου κλπ. τα οποία διέχονται από διαφορετικέ σεισμικέ ζώνε με διαφορετική σεισμικότητα μέσω ενεργών σεισμικών ρηγμάτων σχεδιάζονται λαμβάνοντα υπόψη αυτού του παράγοντε οι οποίοι αυξάνουν σημαντικά το κόστο κατασκευή. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν υπολογίζονται και συγκρίνονται κόστη κατασκευή. Τέλο, με σκοπό να βοηθηθούν οι δικαιούχοι να εξασφαλίσουν χαμηλότερε τιμέ στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων, ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελεκτικό Συνέδριο να παρέχουν περισσότερε πληροφορίε σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργία μια βάση δεδομένων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με στοιχεία κόστους αναμονάδα EU-wide unit cost για τους μηχανικούς που καταρτίζουν εκτιμήσεις για τα νέα έργα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σταματήσω και να σας ευχαριστήσω. Thank you. Then it is uh, no. Ευχαριστώ. Και τώρα οι ευρωβουλευτές μπορούν να αντιδράσουν. Έχω τουλάχιστον δύο στον κατάλογο. Πρώτα η κυρία Παναγιώτοβα. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, να ευχαριστήσω καταρχήν τον εκπρόσωπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την έκθεση που μας παρουσίασε. Είναι μια έκθεση που είναι μια πολύ καλή βάση για τη δουλειά της Επιτροπής μας για τον έλεγχο του προϋπολογισμού και θα ήθελα να συγχαρώ και τον κύριο Σταυρακάκη για τη δουλειά που έκανε να ετοιμάσει την έκθεση. Να αναφέρω τρία βασικά σημεία. Αποτελεσματικότητα, ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, μέσω μιας βάσης δεδομένων σε ευρωπαϊκό δηλαδή επίπεδο και τέλος οι λόγοι για τους οποίους πολλά έργα έχουν καθυστερήσεις. Καταρχάς, υποστηρίζω την προσέγγιση του ελεγκτικού συνεδρίου που δίνει έμφαση στην αποτελεσματικότητα, όχι μόνο στην κανονικότητα των δαπανών, στις μη παρατυπίες δηλαδή. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποιούνται τα χρήματα και τα ωφέλη που έχουν τα έργα αυτά, που απορρέουν από τα έργα αυτά. Είναι πολύ σημαντικό να ποσοτικοποιήσουμε όλα αυτά τα θέματα και την βελτίωση ας πούμε της ασφάλειας των ε, δρόμων. Να δούμε πόσες ζωές σώθηκαν χάρη στους νέους βελτιωμένους δρόμους. Να προσμετρήσουμε δηλαδή τον τρόπο που βελτιώθηκε η ασφάλεια στους δρόμους χάρη στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ψάξουν να βρουν συγκεκριμένους δείκτες για να μετρήσουμε σαφώς τα ωφέλη αυτών των έργων σε εθνικό σε περιφερειακό επίπεδο, βράχει πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Και επίσης συμφωνώ με τις συστάσεις του εισηγητή για αυτή την πιθανή βάση δεδομένων για ανταλλαγή πληροφοριών. Νομίζω ότι θα βοηθήσει αυτούς που οργανώνουν τους διαγωνισμούς για να κάνουν προκαταρτικές εκτιμήσεις για το πώς θα κοστίσει το κάθε τι. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε αποτελεσματικοί όταν δημιουργούμε τις δομές χάρη στην ανταλλαγή των πληροφοριών. Έχουμε ακόμα μία έκθεση, σας το υπενθυμίζω και έχουμε και άλλους ομιλητές. Έτσι έχω και κάποιες άλλες συστάσεις να κάνω. Εν συνεχεία, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά τους λόγους για τις καθυστερήσεις που έχουν κάποια έργα και να δούμε σε ποιο βαθμό αυτές οι καθυστερήσεις ε, οφείλονται στο α ή στο β. Γιατί έχουμε συγκεκριμένα συγκεκριμένες καθυστερήσεις σε κράτη-μέλη λόγω ας πούμε κακού προγραμματισμού ή άλλων προβλημάτων. Μερικές φορές βέβαια οι καθυστερήσεις οφείλονται και σε απρόβλεπτες ιστορίες όπως παραδείγματο χάρη προσπελασιμότητα της περιοχής, αρχαιολογικά ευρήματα κτλ. Ακόμα είμαστε στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να συμπεριληφθεί αυτό το κείμενο στην έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γιάλα Σέντερ. Σύντομα θα ήθελα να σας παρακαλέσω. Ευχαριστώ τον εισηγητή για τις εξηγήσει του. Αυτό μου φαίνεται εντυπωσιακό, συγκλονιστικό θα έλεγα, είναι το θέμα του κόστους. Το είδαμε. Είδαμε ότι τετραπλασιάζεται στην ε, Ισπανία το, το κόστος χωρίς να υπάρχει εξήγηση. Κοίταξε λίγο την έκθεση. Φαντάζομαι ότι ο υπεύθυνο του ελεκτικού συνεδρίου κοίταξε πολύ λεπτομερό την έκθεση. Μπορούμε να συγκρίνουμε βέβαια τους τιμούς στην Ισπανία και στην Γερμανία, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε και άλλα πράγματα. Πρέπει να καταλάβουμε πού οφείλονται αυτές οι τεράστιες διαφορές. Με βάση το ελεγκτικό συνέδριο και την έκθεσή του υπάρχουν τρεις τρόποι αξιολόγησης του κόστους. Έχεις ε, το συνολικό κόστος της κατασκευής, Πρέπει να δούμε κατά πόσον χτίζονται χτί, ε, γέφυρες, ε, σύραγγες, ε, περιβαλλοντικά προβλήματα. Αλλά δεν μας ανέφερε τίποτα για όλα αυτά το ελεκτικό συνέδριο. Το να χτίζουμε στην Ισπανία δεν είναι το ίδιο με το να χτίζουμε οτιδήποτε στη Γερμανία. Το κόστος ανά χιλιόμετρο είναι πολύ διαφορετικό σε εμά. Θα ήθελα να μου δοθεί μια εξήγηση για αυτές τις τρομερές διαφορές κόστους. Λέτε ότι στην Ισπανία είναι τέσσερις φορές πιο ακριβό το κόστος, αλλά δεν λέτε γιατί και τι γίνεται και με το κόστος της κρίσης. Πώς το λαμβάνει υπόψη το ελεγκτικό συνέδριο. Εσείς λέτε το κόστος ε, στην Ισπανία είναι τετραπλάσιο. Αυτός ο υπολογισμός βασίζεται στην ε, μέση κυκλοφορία. Από το 2008 μειώθηκε η κυκλοφορία σε σχέση με τα νούμερα που υπάρχουν εδώ. Κύριε Βάιζενμπεργκ, θα ήθελα να μας δώσετε όλα τα στοιχεία που έχετε, όχι αποσπασματικά, όχι λίγα από εδώ, λίγα από εκεί. Σας παρακαλώ λοιπόν να μας δώσετε μια πιο συνολική εικόνα και να μας δώσετε και κάποιες διευκρινήσεις για το πώς συνυπολογίζεται το κόστος ε, της κρίσης στην Ισπανία, Γερμανία και Πολωνία. Το κόστος ε, οικοδόμησης δρόμων στην Ισπανία, γιατί είναι τετραπλάσιο. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε μια ορεινή χώρα, Φερρυπίν, και πρέπει να περάσουμε μέσα από τα βουνά και αυτό κοστίζει. Πρόεδρος, λόγω του χρόνου και επειδή ξοδέψαμε 20 λεφτά ήδη σε αυτή την έκθεση και έχουμε ακόμα μία έκθεση στην ημερησία διάταξη και νομίζω ότι είναι δίκαιο όλος, όλοι να έχουν λίγο χρόνο να μιλήσουν. Θα ήθελα λοιπόν η Αγέλα, κυρία Γιάλα Σέντερ να ε, δει διμερός τον εκπρόσωπο του Ελληνικού Συνεδρίου και ελπίζω να πάρει τις απαντήσεις που θέλει. Ούτως ώστε να σταματήσει εδώ αυτή η συζήτηση. Και ο εισηγητής να κάνει τα τελικά του συμπεράσματα. Είσαστε εντάξει, δεν θέλετε να μιλήσετε. Συμφωνείτε όλοι. Δεν θέλω να γνωρίσω και την Κομισιόν φυσικά, γιατί έχουν και τον τελικό λόγο για αυτά τα θέματα. Ξέρω ότι η Κομισιόν είναι πάντα λακωνική και ελπίζω σήμερα λοιπόν να είναι εξίσου λακωνική με τη φήμη της τουλάχιστον. Ευχαριστώ. Καλωσορίζουμε, Πρόεδρε, την έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου. Μιλάει για ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο εξετάσαμε και εμείς επί χρόνια. Ε, ευχαριστούμε και για τα συμπεράσματα της Επιτροπής σας. Ε, το πρώτο σημαντικό σημείο είναι ότι γενικά συμφωνούμε με τα πορίσματα και με τις συστάσεις. Για πολλές από τις συστάσεις είμαστε σε διαδικασία μετρήσεων και για την επόμενη περίοδο του προγραμματισμού προσπαθούμε εκεί να εστιάσουμε τώρα, γιατί αυτό είναι ο πιο σημαντικός τρόπος για να προχωρήσουμε. Πρέπει δηλαδή αυτές τις ε, ελλείψεις να τις ε, αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Επίσης, έχουμε διάφορα εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε για να διορθώσουμε κάποια από τα προβλήματα. Καταρχάς, θα πρέπει να είμαστε πιο στρατηγικοί. Να δούμε δηλαδή τι δρόμους θα επιλέξουμε για υποστήριξη. Θα θέλαμε δηλαδή καταρχάς να έχουμε ε, μια στρατηγική θεώρηση, εθνικά προγράμματα και να έχουμε ένα συνολικό πλαίσιο όλων των, προγραμμάτων δηλαδή, που θα υποστηριχθούν με τοπικά και ευρωπαϊκά κονδύλια. Ε, και εθνικά φυσικά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό σημείο για το μέλλον. Κάτι άλλο σημαντικό, στην ε, εξάντε αιρεσιμότητα ε, βάζουμε, δίνουμε εστίαση, βάζουμε εστίαση και στις δημόσιες προμήθειες, γιατί υπάρχουν κάποια λάθη στους διαγωνισμούς. Ορισμένα από τα προβλήματα οφείλονται στην δημοσίευση. Ε, υπάρχει αυτή η εκ των προτέρων ρεσιμότητα. Το θέμα δεν είναι πώς εφαρμόζονται αυτά τα προγράμματα, το θέμα είναι να υπάρχει διαφάνεια, κατάρτιση. Αυτά είναι συγκεκριμένα μέτρα για να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να υπερβούν τις αδυναμίες για τη διαχείριση των έργων. Διοικητική ικανότητα, πώς συντάσσεται το, τα, έγγραφα, ε, πώς εφαρμόζεται ένα περίπλοκο έργο. Γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτά είναι περίπλοκα έργα. Στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού, λοιπόν, τι θα κάνουμε. Θα δουλέψουμε με δείκτες, θα υπάρχει ένα πλαίσιο επιδόσεων και θα εξασφαλίσουμε ότι αν κάποια από τα αποτελέσματα δεν έχουν υλοποιηθεί, θα περάσουμε στην αναστολή της χρηματοδότησης. Επομένως, ε, συνδέομαστε περισσότερο ανάμεσα στους στόχους και στα αποτελέσματα. Υπάρχει μεγαλύτερη σύνδεση, δηλαδή, ανάμεσα στους στόχους και στα αποτελέσματα των έργων. Και άλλο σημαντικό στοιχείο. Έχουμε διάφορα μέτρα, λοιπόν. Φυσικά θα συνεργαστούμε με το ελεγκτικό συνέδριο σας ευχαριστώ ακόμα μια φορά για την έκθεση και ευχαριστώ και την Επιτροπή σας για τα συμπεράσματά της. Χαιρόμαστε που ήδη το ελεγκτικό συνέδριο συνέχισε, ε, συνένεσε με αυτά που είπε η Κομισιόν. Πάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ειδική έκθεση υπαριθμών 6. Τα κράτη-μέλη και Κομισιόν έχουν πετύχει αυτά που έπρεπε με βάση τα λεφτά που δόθηκαν στα μέτρα ε, διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας. Ο κύριος ευχαριστώ. Να σας πω γρήγορα το τι ελέγξαμε και το τι βρήκαμε. Όπως ξέρετε, πάρα πολλές ε, περιοχές ε, της Υπέθρου έχουν έλλειψη οικονομικών ευκαιριών αλλά και χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού. Μπορούν λοιπόν οι επιδοτήσεις ε, να συνεισφέρουν σε αυτό. Αυτή τη στιγμή η τωρινή πολιτική περιλαμβάνει τρία μέτρα που ακριβώς στοχεύουν στην διαφοροποίηση της ε, οικονομίας της υπαίθρου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει 5 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2007-2013 και αυτό συμπληρώνεται με εθνικές δαπάνες και έτσι φτάνουμε σε ένα σύνολο 7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το οποίο βρήκαμε λοιπόν είναι το εξή. Πρώτον, τα κράτη-μέλη δεν κατέδειξαν σαφώς ανάγκη για αυτά τα μέτρα και δεν έχουν καθορίσει γιατί και πώς η δημόσια παρέμβαση σε μη γεωργικές δραστηριότητες μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα ανάπτυξης και απασχόλησης. Έτσι, ουσιαστικά οποιοδήποτε έργο μπορεί να ενταχθεί στους στόχους αυτούς. Κατά την ε, άποψη του Ενεκτικού Συνεδρίου, η Κομισιόν δεν θα έπρεπε να έχει εγκρίνει προγράμματα που δεν αποδείκνυαν σαφώς την ανάγκη δαπάνης και ποια είναι τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Οι στόχοι αυτοί συνδυάστηκαν με δύο κριτήρια επιλεξιμότητας και συστήματα τα οποία είτε δεν είχαν νόημα είτε δεν εφαρμόστηκαν καθόλου. Άρα επιλέχθηκαν όσο δυνατόν περισσότερα επιλέξιμα έργα με τους ε, πόρους που υπήρχαν, ανεξαρτήτως του πώς αξιολογήθηκαν όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους. Τέλος, όταν ε, ήταν δεσμευμένη η χρηματοδότηση, έπρεπε να επιλεγούν τα λεγόμενα καλύτερα έργα. Δεύτερον, τα κράτη-μέλη δεν διοχέτευσαν συστηματικά την χρηματοδότηση εκεί όπου υπήρχε σαφής ανάγκη για ε, χρηματοδότηση του δημοσίου. Παραδείγματο χάρη 35 από τα 57 έργα θα είχαν γίνει ούτω ή άλλω και χωρί χρηματοδότηση του δημοσίου. Σχεδόν στα μισά κρίναμε πω η επένδυση είχε ήδη ξεκινήσει και σε μια περίπτωση και κιόλα ολοκληρωθεί πριν ενταχθεί στο πρόγραμμα. Πρόκειται βεβαίω ξεκάθαρα για μια περίπτωση φύρας. βεβαίως έτσι βελτιώθηκε η θέση του δικαιούχου αλλά εις βάρος ενός ανταγωνιστή χωρίς ε, κάποιο όφελος στην πραγματική οικονομία. Τέλος δεν υπήρχαν αξιόπιστες πληροφορίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των μέτρων. Ξέρετε κύριε Πρόεδρε πώς τα έχουμε ξαναπεί αυτά και σε προηγούμενες εκθέσεις. Ε, η τελευταία ήταν μόλις πριν από δύο εβδομάδες. Τα στην έκθεση Κάντενμπαχ. Τέλος, κύριες Πρόεδρε, θα ήθελα να προσθέσω πως ακόμα και αν έχει συμφωνηθεί σε πολιτικό επίπεδο στόχος αυτός, μπορούμε να λάβουμε υπόψη τα συμπεράσματα του ελέγχου στις πράξεις κατεξιοδότηση για να προετοιμαστούμε για το 2014. Επίσης, ο κανονισμός αντιμετωπίζει κάποια ζητήματα, όπως η έλλειψη ανάλυσης αναγκών ή τα κριτήρια επιλογής έργων, οι πράξεις κατά εξοδότηση μπορούσαν να λάβουν υπόψη κάποια στοιχεία που αναφέρει η τα κριτηρια επιλογης εργων η πραξη κατα εξοδοτηση μπορουσαν να λαβουν υποψη καποια στοιχεια που αναφερει η εκθεση Π.χ. η διαδικασία έγκρισης της Κομισιόν που εμείς θεωρούμε πως θα πρέπει να κάνει μια πιο κριτική αξιολόγηση των αιτιολογήσεων των μελών. Άλλες πτυχές που θα ήθελε να δει το ελεγκτικό συνεδρίο είναι κριτήρια επιλογής τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη την ποιότητα των έργων και ενός ε, συστήματος βαθμολογίας και η δυνατότητα της Κομισιόν να επαληθεύει την εφαρμογή από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Κυρία Κάντεμπαχ, θα ήθελε να πει κάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γιάν Κίνστ. Και είμαι μέλος επίσης ε, και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Γεωργίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Και οι τρεις αυτές ε, επιτροπές βεβαίως ε, έχουν το πρόβλημα της κατανομής των μέσων και της χρήσης των κονδυλίων. Και βεβαίως υπάρχει και το ζήτημα της διαδικασίας τοποθέτησης του Κοινοβουλίου. Πάρα πολλά ζητήματα δεν έχουν ακόμα θυγεί γιατί θεωρώ πως θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στις τροπολογίες. Ε, δηλαδή εκεί όπου μιλάμε για ποιότητα ζωής στην Ήπεθρο, ανάπτυξη και σε επαγγέλματα και σε επαγγελματικές ομάδες εκτός της γεωργίας και κυρίως, και εδώ πέρα είναι και ένας από τους στόχους, για να παραμείνουν οι νέοι στην Ήπεθρο. Δεν επαρκεί ε, δηλαδή να υπάρχουν ε, μόνο οι επιδοτήσεις αλλά και οι αναγκαίες ε, υποδομές, γιατροί, παιδικοί σταθμοί και λοιπές κοινωνικές υπηρεσίες. Πρέπει εδώ πέρα λοιπόν να δούμε τι θα πει το ελεγκτικό συνέδριο, να το λάβουμε υπόψη στην ε, επόμενη έκθεση για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην ε, Ήπεθρο. Τέλος, ε, θεωρώ πως κάποια από αυτά τα οποία αναφέρθηκαν μπορούν να αλλάξουν στην επόμενη προγραμματική περίοδο από το 2014 γιατί ούτως ή άλλως η ανάπτυξη της Πέθρου θα έχει τελείως διαφορετική μορφή και ε, νομίζω είναι η δική μας η αποστολή μαζί με τα κράτη-μέλη να δούμε ποια θα είναι η εφαρμογή της πολιτικής αυτής στην Ήπεθρο σύμφωνα με τις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Γιατί νομίζω επαφίεται και στα κράτη-μέλη το πώς θα εφαρμόσουν το πλαίσιο αυτό Ήδη από την επιλογή των έργων θα πρέπει να υπάρξει μια κρίση εξ για το εάν τα έργα αυτά έχουν μια πιθανότητα να εκπληρώσουν τους στόχους που υποτίθεται ότι έχουμε θέσει. Σας ευχαριστώ. Τώρα... Οι ευρωβουλευτές μπορούν να αντιδράσουν. Έχετε το λόγο. Ο κύριος Ρούμπιχ. Να ευχαριστήσω την κυρία Κάντεμπαχ είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό για το μέλλον, το μέλλον μας. Είναι θέμα του πώς θα διασφαλιστεί η ανάπτυξη. Δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχουν σαφή κριτήρια ενίσχυσης. Οπότε λογικό θα ήταν νομίζω στο μέλλον να ενισχυθεί η αυτοαπασχόληση, οι μικρές επιχειρήσεις μέχρι 10 ε, υπαλλήλου. Ε, εδώ πέρα νομίζω μπορούμε να έχουμε το μεγαλύτερο αποτέλεσμα σε μειονεκτικές περιοχές και θεωρώ τέλος πως η ενίσχυση αυτών των δραστηριοτήτων στις περιφέρειες πρέπει να βρεθεί στο προσκήνιο. Η απασχόληση ε, πρέπει να έχει προτεραιότητα. Δεν θα μπω τώρα στις λεπτομέρειες. Αυτό είναι το αποφασιστικό. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Δεν θέλει κανένα άλλο το λόγο που θέλει να αντιδράσει. Να μην ξεχάσω και την Κομισιόν. Ο κύριος Ντεσόζα, ο παλιός μου φίλος είναι εδώ, του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ το συνέδριο και τον εισηγητή για τις παρατηρήσεις και συστάσεις. Να τονίσω ότι η ισχύουσα νομοθεσία καλύπτει όχι μόνο την εφαρμογή, αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής στις αγροτικές περιοχές και την διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων. Η Κομισιόν θεωρεί ότι πολλές από τις συστάσεις του συνεδρίου απευθύνονται στα κράτη-μέλη, φερειπίν σε ό,τι αφορά την επιλογή των βιώσιμων ε, έργων ή αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου. Η αρχή της επικουρικότητας επίσης ε, και περιγραφές για τα κράτη-μέλη και τις περιοχές ε, των μέτρων διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας. Φυσικά υπάρχουν, ε, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και αυτή η βελτίωση μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Με την ενίσχυση στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού της στρατηγικής προσέγγισης, πιο αποτελεσματική και πολιτική ανάπτυξη της υπαίθρου. Επιλεγμένα μέτρα που θα βασίζονται σε ε, λογική ε, πολιτική παρέμβαση με σωστή αξιολόγηση. Όταν τα προτινόμενα προγράμματα δεν ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της παρέμβασης και δεν έχουν συγκεκριμένους στόχους, τότε η Κομισιόν θα τα εγκρίνει. Περαιτέρω βελτιώσεις είναι δυνατές ό,τι αφορά την ε, εφαρμογή και θα ήθελα να τονίσω ότι θα έχουμε μια νέα προσέγγιση που θα βασίζεται στα αποτελέσματα που υποστηρίζει την πολιτική ανάπτυξη υπαίθρου. Ε, αυτά που είπε το ελεγκτικό συνεδρίο συγχωνεύονται σε ένα πλαίσιο με καλύτερη εστίωση για την, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τη βελτίωσή τους και με στόχο τη μείωση του γραφειοκρατικού άχθους. Η Κομισιόν συμφωνεί με το συνέδριο ότι το σύστημα επιλογής των έργων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ποιότητα των έργων αυτών και να χρησιμοποιεί ένα σύστημα βαθμολόγησής τους. Αυτά τα αποτελέσματα θα ενισχυθούν. Ε, δίνουμε οδηγίες στα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τα κριτήρια επιλογής και τις συνθήκες επιλεξιμότητας για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού για να βελτιώσουμε αυτά τα σημεία. Επίσης, οι συζητήσεις συνεχίζονται σε ό,τι αφορά το ποσοστό μετατόπισης. Θα έχουμε ένα πιο συγκεκριμένο ε, πλαίσιο ό,τι αφορά τη φύρα. Επίσης, να τονίσω τα εξή σημεία. Η επιλεξιμότητα των δαπανών στο ταμείο μας ε, γίνεται δεκτή αν αφορά επιχειρήσεις που που ελέγχουν οι διαχειριστικές αρχές με βάση τις αρχές της επιλογής των έργων. Η επιλεξιμότητα των δαπανών που γίνεται θα πρέπει να συνοδεύεται με αίτηση προς αρμόδιες αρχές σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις που εντάσσονται ε, στα πλαίσια του άρθρου 42 της Συνθήκης. Η Κομισιόν έχει ε, μέτρα για να βελτιώσει περαιτέρω την πολιτική και την εφαρμογή της. Ε, καταρχάς, ελεγξιμότητα και αξιοπιστία των μέτρων τη στιγμή που δημιουργούνται. Σε ό,τι αφορά το εύλογο κόστος, οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν ε, έγγραφα για να ξεκινήσουν α, τις επιχειρήσεις και το, η τελευταία δόση θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο εφαρμόζονται επιτυχώς αυτά τα προγράμματα. Επίσης, οι επενδύσεις σε αυτές τις περιοχές θα είναι επιλέξιμες αν είναι σύμμορφες με τα σχέδια ανάπτυξης ε, των δήμων και κοινοτήτων, ε, αν υπάρχουν αυτά τα σχέδια, ούτως ώστε να είμαστε και συνεπείς με οποιαδήποτε τοπική στρατηγική ανάπτυξης. Για την παρακολούθηση και αξιολόγηση θα χτενίσουμε το πλαίσιο που υπάρχει ήδη για την αξιολόγηση και θα εφαρμόσουμε ένα νέο πλαίσιο το οποίο θα είναι πιο απλό. Έτσι θα αξιολογούμε την πρόοδο και την, ε, της εφαρμογής με βάση κοινού ε, δείκτες για τις προτεραιότητες σε επιλεγμένες περιοχές ε, των έργων. Η Κομισιόν θεωρεί ότι οι προβλεπόμενες πρωτοβουλίες θα λάβουν υπόψη τις συστάσεις του συνεδρίου και ούτως ή άλλως δεν ξεχνάμε ότι όπως είπε και ο εισηγητής δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι ο στόχος μας είναι η βελτίωση της ζωής των ανθρώπων στην Ήπεθρο και η ενθάρρυνση της, των ποικιλόμορφων οικονομικών δραστηριοτήτων στις περιοχές αυτές. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος της συζήτησης. Συνένεση υπάρχει μεταξύ όλων των ομιλητών για τους δείκτες και Δεύτερον, ότι κυρίω οι εθνικέ κυβερνήσει πρέπει να βελτιώσουν την ε, κατάσταση, κυρίως. Με αυτά τα συμπεράσματα σταματούμε εδώ τη συνεδρίαση και θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9 στην ίδια αίθουσα. Γεια σας. On n'a pas eu